Good morning, everybody, dear colleagues. Καλημέρα, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Θα ομιλήσω την Ισπανική, μπορείτε να φορέσετε τα ακουστικά σας. Buenos Σας καλημερίζω λοιπόν για μια ακόμη φορά λέει η Πρόεδρος εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Σας καλωσορίζω στην αίθουσα αυτή. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σε αυτό το Gender Summit όπως λέμε Ελπίζω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα έχει ενδιαφέρον για όλους. Τη στιγμή κατά την οποία οι τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν, δεν μπορεί να μας κάνουν να αγνοήσουμε ορισμένα βασικά θέματα τα οποία παραμένουν διαχρονικά Και ακριβώς αυτή είναι, αυτός είναι και ο προσανατολισμός της δράσης μας και σε πολιτικό επίπεδο και σε διερευνητικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται έτσι ώστε να βελτιώσουν την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και την ευημερία των μεν και των δε ποιότητα λοιπόν της καινοτομίας μέσα από την ισότητα. Θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε εξαιρετικούς ομιλητές που θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους και τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ, τους αγαπητούς ομιλητές. Εμείς συζητάμε μια έκθεση πρωτοβουλίας στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή για την πολιτική ισότητα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Και προσπαθούμε στα πλαίσια των στόχων που έχουμε θέσει σαν Επιτροπή να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε τον εγκάρσιο χαρακτήρα της ισότητας των φύλων να την εντάξουμε σε όλες τις πολιτικές μας είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης στον τομέα της καινοτομίας και στον τομέα της έρευνας. Θα πρέπει να εντάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα τον καθολικό της προβληματικής του φύλου έτσι ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να καλύψουμε τις ανάγκες του μισού πληθυσμού της Ευρώπης και του κόσμου. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ για να συναντηθούμε Ελπίζω ότι με τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουμε στο τέλος της συνεδρίασης να έχουμε περισσότερα επιχειρήματα, πιο ξεκάθαρες θέσεις που θα ωφελήσουν τις εργασίες των ΜΕ και των ΔΕ. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να δώσω το λόγο στον κύριο Μάριο Πίντο, επίτιμο συμπρόεδρο αυτής της συνάντησης, Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα. Θα μοιραστούμε την Προεδρία λοιπόν σήμερα. Κύριε Πίντο έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ. Είναι live stream Ε, μετάδοση, αναμετάδοση στο διαδίκτυο γιατί αναφέρεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μετάφραση και δεν ε, αναμεταδίδεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σαν γλώσσες εργασίας όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής <clears throat> Ένωσης. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την εξαίρετη προσφορά των διερμηνέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με στόχο να μπορέσει ο καθένας από εσά να εκφραστεί στη μητρική του γλώσσα. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι και αλλιώ ο κύριος Πίντο θα μπορέσει να ομιλήσει ε, με την γλώσσα την οποία, στην γλώσσα την οποία αυτός θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμη. Άλλωστε ο καθένας από εμά έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί καθημερινά την γλώσσα που επιθυμεί. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση του Καναδά. Θα ήθελα να κάνω κάποιε προκατακτικέ ε, παρατηρήσει προτού περάσουμε στην ε, ε, πρώτη σύνοδο. Ο ρόλος επιστήμη και της τεχνολογίας εν γέννη. Περί τίνο πρόκειται άνθρωποι, διάλογος, επαφές, ανταλλαγές σε σχέση με τις γνώσεις που έχουμε. Όμως η επιστήμη δεν είναι μόνο για την ελίτ, ε, σε την Όλοι ε, θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να υποφεληθούν από τις νέες γνώσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις των επιστήμων του, του, του, επιστημονικού προσωπικού ως ε, μόχλευση ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε τα επιστημονικά προγράμματα και τα αποτελέσματα της έρευνας ανά τον κόσμο ούτως ώστε όλοι να αποκομίσουν ωφέλη από την έρευνα θα πρέπει να προβληματιστούμε πώς το περιβάλλον της έρευνας θα μπορούσε να αποτυπώνει γενικότερα τον κοινωνικό ιστό. Ε, εάν βλέπουμε νέες απόψεις, νέες εμπνεύσεις και επικοινομορφία από απόψεων θα πρέπει να ε, εμπλέκονται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορούμε πλέον να παραγνωρίζουμε περιθωριοποιημένες μέχρι τούδε κοινωνικές ομάδες στον ακαδημαϊκό κόσμο. Παραδείγματος χαρή αυτόχθονες στον Καναδά. Ε, χρησιμοποιούμε ορασία από δύο διαφορετικά μάτια, έτσι ονομάζεται, για να έχουμε δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες και να αναπτύξουμε έτσι μια ολιστική κοσμοθεωρία. Αυτή ε, τη θεώρηση των πραγμάτων επιδιώκουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, γενικότερα και ειδικότερα στον τομέα της έρευνας, ε, διότι είναι ένα τόσο πολύτιμο εργαλείο για να επιτύχουμε την ισότητα των ευκαιριών. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να σας ξαναδώσω το λόγο Πρόεδρε μετά από αυτά τα σύντομα σχόλια. Χαίρομαι ιδιαίτερος που συμμετέχω σε αυτό τον διάλογο για την πολιτική. Θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ε, κοινωνικό ευζήν μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίντο. Ε, δίκιο έχετε όταν λέτε πως... Ε, όταν λέτε πως ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως είναι ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό και αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για ε, να σημειώσουμε προόδο στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γι' αυτό και για άλλα ζητήματα πιστεύω ε, η πρωινή μας σύνοδος θα είναι πάρα πολύ ε, καρποφόρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Grace Ναλέντι Μαντίσα Παντόρ, που είναι η Υπουργό τη Νοτιού για την Επιστήμη και την Τεχνολογία. σας ευχαριστούμε που κάνατε όλο αυτό το δρόμο για να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να ε, σας προσφωνήσω σε αυτή την τόσο σημαντική σύνοδο. Ε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους σας για την πρόσκληση που μου απίφθηναν. Θα ήθελα προς αξιότιμους καλεσμένους να υπενθυμίσω ότι εδώ και 22 χρόνια μόνο χαιρόμαστε και εποφελούμαστε από τη δημοκρατία στη Νότια Αφρική και αρχίσαμε να κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται για να επανορθώσουμε όλες τις ανισορροπίες που ήταν η απόρρια της ιστορίας μας, της αποξένωσης και του αποκλεισμού. Έτσι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αποκατασταθούν και στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στο θέμα της ισότητας των δύο φίλων. Η πορεία του εκδημοκρατισμού της ανώτερης παιδείας άρχισε ιδιαίτερο στο 1994 με την ε, έλευση της δημοκρατίας. Αυτή η περίοδος αλλαγών ε, συμπεριλαμβάνει και τον αγώνα κατά ε, της διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω εθνότητας ή λόγω φύλου. Και ε, είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να αντιμετωπίσουμε την αποξένωση, τη συμμετοχή των ε, ε, μαύρων στην κοινωνία, τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα διακριτικών μεταχειρήσεων και αποκλεισμών που, και σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την κυβερνητική μας πολιτική. Στα 22 χρόνια εκδημοκρατισμού ε, σημειώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος ε, κυρίως ε, στον τομέα της ανώτερης παιδείας. Όμως υπολείπονται σημαντικότερες προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Συνοψίζοντα, μπορώ να σα πω ότι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά τη χώρα μα, κυρίω στον τομέα τη παιδεία σε ανώτερε βαθμίδε, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών είναι νέοι μαύροι, ε, ε, γυναίκες και άντρες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των γυναικών στην παιδεία ε, στη Νότια Αφρική, στις ανώτερες βαθμίδες, έχει γίνει σοβαρότατη επένδυση στους νέους και στην πρόσβαση των γυναικών σε νέες ευκαιρίες. Όμως, παρότι διαπιστώνουν τις ανώτερες βαθμίδες παρουσία των γυναικών. Παρότι υπάρχει ισότητα υπέρ ε, των γυναικών, ε, δυστυχώς γέρνει η πλάστιγκα στους κρατικούς θεσμούς προς τους άντρες. Για τις ε, σταδιοδρομίες στον τομέα της επιστήμης, για την διαδικασία διδακτορικών. 58% των γυναικών φτάνουν ε, στο επίπεδο προδιπλώματος ένα τμήμα αυτό των γυναικών ε, συνεχίζουν σε διπλώματα, αλλά σε επίπεδο μάστερ εγκαταλείπουν πάρα πολλές γυναίκες στις σπουδές και ακόμη περισσότερες σε επίπεδο διδακτορικού. Τέτοια ζητήματα θα πρέπει να ρυθμίσουμε, ούτω ώστε να μεγενθύνουμε την επιρροή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έχουμε <clears throat> αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες ε, για να ρυθμίσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Ε, το πρόγραμμα του ΤΟΥΚΑ, παραδείγματος χαρητή, σημαίνει «φροντίζω». Ε, υπάρχουν τρεις πορείες επιταχυμένες για τις γυναίκες, για το διδακτορικό, μετά-διδακτορικό και για ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα. Χρηματοδοτείται <clears throat> από την κυβέρνηση και παρέχει στήριξη στις γυναίκες. Δεύτερη πρωτοβουλία είναι η συγκρότηση κέντρων αριστείας με ε, υπότροφους και ερευνητές ε, καταξιωμένους που δύναται να έχουν ηγετικό ρόλο στα κέντρα αριστείας 16 ε, το αριθμό μέχρι στιγμής όμως ένα μόνο ηγείται σε ένα μόνο ηγείται ε, γυναίκα, στα υπόλοιπα 15 είναι άντρες οι διευθυντές. Τρίτο μοντέλο παρέμβασης, το από τον Καναδά αυτό, είναι μία ε, πρωτοβουλία ερευνητική για τις έδρες, ε, για τους διδακτορικούς φοιτητές και για τους ερευνητές. Μέχρι το 2015 είχαμε 157 έδρες και η μισή που έκαναν διδακτορικό ήταν άντρες και οι άλλες μισές γυναίκες. Όμως από τις 157 έδρες μόνο οι πέντε ήταν, ε, ε, αποδόθηκαν σε γυναίκες. Ε, το βρήκα Λίαν ε, απογοητευτικό όταν είδα τις στατιστικές ε, και για την πολιτική, επειδή είχα την δυνατότητα να δράσω, το 2015 αποφάσισα ότι εφ' ε οι νέες έδρες για το 2015 θα πρέπει να ε, καταληφθούν από γυναίκες υποψήφιους ε, και με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι δεν έχουμε τόσες γυναίκες επιστήμονες στη Νότια Αφρική. Από στις 40 έδρες ε, οι επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση, όταν ανοίξαμε την πρόσκληση υποβολής προσφορών και αναφέραμε ότι οι γυναίκες θα είχαν προβάδισμα, ήρθαν όμως 63 αιτήσει ε, από γυναίκες που ε, είχαν κάθε δεξιότητα ε, που απαιτείται για να καταλάβουν αυτές τις έδρες. 42 ε, από τις νέες έδρες λοιπόν καταλήφθησαν από γυναίκες και ως policy maker έμαθα ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα και ποιο ήταν αυτό το δίδαγμα ότι η ριζοσπαστική παρέμβαση και η πολιτική δράση είναι προαπαιτούμενα για να επέλθει η αλλαγή στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το ΣΑΡΚΙ 42 με αυτές τις έδρες αλλάζει τις ε, στατιστικές. Ε, μόνο ένας από τους τρεις επιστήμονες είναι γυναίκες ε, και είναι νεότεροι και έχει λιγότερες δεξιότητες σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους. Υπολείπεται πολύ μεγάλο έργο. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για να υποστηρίξουμε και να αναγνωριστεί ο ρόλος των γυναικών στην επιστήμη, διότι χωρίς αυτές δεν θα επέλθει σημαντική αλλαγή. Ε, την πρόσβαση για τις επιστήμονες ε, θα είναι ένα βασικό στοιχείο τόσο ώστε σε ε, τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία και και η παράλληλη οικονομία ε, θα μπορέσουν ως νέοι τομείς έρευνας ε, να χαρακτηριστούν από έντονη παρουσία των γυναικών. Ε, ως ε, νεόφυτες ε, σε αυτούς τους επιστημονικούς τομείς ε, θα μπορέσουν να καταξιωθούν όπως και οι άντρες επιστήμονες έχοντας έτσι τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις σε, αυτές του σε αυτούς τους σημαντικούς θεσμούς που υποστηρίζει η κυβέρνησή μας. Νομίζω ότι σας έδωσα τώρα κάποιες ενδείξεις για την κατάσταση στην Νότια Αφρική. Έχει σημειωθεί η προόδος, έχουμε δημιουργήσει πρόσφορο περιβάλλον για την πρόθεση του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη, τεχνολογία και στον τομέα της καινοτομίας όμως έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Εν κατακλείδη θα ήθελα να ασχοληθώ γενικότερα με την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε δισεκατομμύρια πληθυσμό και ε, έχουμε και την ταχύτερη ανάπτυξη στον κόσμο. Ε, επιδιώκουμε ε, μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών που εξάγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε η ανάπτυξη να μην αποκλείει κανέναν ναι, και τα ωφέλη να ε, να, μοιράζονται σε όλους ε, στην Αφρική ε, και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το επιτύχουμε είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, ούτως ώστε σε ευρύτερο αριθμό τομέων της αφρικανικής οικονομίας να υπάρχουν αξιοπρεπείς θέσει εργασίας, να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας με αποφασιστικότητα ούτω ώστε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε αυτές τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, να προωθήσουμε βιομηχανίες όπως η γεωργία, ο κατασκευαστικό ε, τομέα τουρισμό ε, ε, τουρισμός, μικρές που δημιουργούν πολλέ θέσει εργασία η μεταποίηση επίσης, οικονομικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, και ε, επιχειρηματικές υπηρεσίες. Όλοι αυτοί οι τομείς τι χρειάζονται, δεξιότητες, επιστήμη και ε, καινοτομία. Χρειαζόμαστε τις γυναίκες της Αφρικής. Η βελτιστοποίηση της παρουσίας τους και τη συμμετοχή τους στην οικονομία, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και στην μεγέθυνση των γνώσεων που επιτρέπουν η οικονομική ανάπτυξη είναι κάτι απαραίτητο. Η ισότητα των ευκαιριών στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι ένα θέμα που πρέπει τα αντιμετωπίσουμε. Για μας τους policy makers ε, είναι σοβαρότατη η πρόκληση, το ίδιο για τις κυβερνήσεις, για τα κοινοβούλια των χρόνων. Πιστεύουμε ότι στον τομέα της έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας είναι κύριος ο ρόλος των γυναικών, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εθνών κινητήριος δύναμη για την ε, καινοτομία στην Αφρικανική Ήπειρο είναι κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο πέραν της Αφρικής, ε, διότι θα αλλάξει ο τρόπος σκέψης, ο κόσμος θεώρηση των πραγμάτων, πώς αντιμετωπίζουμε ε, την ε, επιστήμη και την τεχνολογία. Η κοινωνική μετεξέλιξη που μπορεί να εδραστεί στην επιστήμη και την τεχνολογία, την καινοτομία, θα αλλάξει την θεώρηση που έχουμε για κάθε επιμέρους τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Είμαστε απολύτως αποφασμένοι να εθαρρύνουμε τις επιστήμονες να εργαστούν στην ε, ε, Αφρική. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνούμε, όπως και στη Νότια Αφρική, να επιλέγουμε τους winners, αυτούς που είναι φτιαγμένοι για την επιτυχία, ε, που θα αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ε, για τους οποίους είμαστε σίγουροι θα καταλάβουν τις ε, υψηλότερες θέσεις και θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή την προσπάθεια πρόθεση επιστήμης τεχνολογίας και της καινοτομίας. Πρόεδρε, έχουμε σημειώσει πρόοδο στη χώρα μου, στη Νότια Αφρική. Είμαστε στις απαρχές της επιτυχημένης πορείας. Σε πολλές χώρες επιδιώκεται να αυξηθούν οι επενδύσεις. Σε αυτούς τους τρεις τομείς, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, για να φτάσουν όμως οι γυναίκες στα ανώτατα κλιμάκια, ε, θα πρέπει να κάνουμε πολλά ε, περισσότερα και ελπίζω μέσα από αυτή τη σύντομη συμβολή σήμερα το πρωί θα σας ενθαρρύνω και εσάς ε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιδιώξετε το ίδιο στενό στενότερες εταιρικές σχέσεις ε, με γυναίκες ε, που καταρτίζουν πολιτική στην Αφρικανική Ήπειρο, ώστε από κοινού να αλλάξουμε ε, τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν οι γυναίκες όχι μόνο στην Αφρική αλλά ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señora. Ευχαριστώ πολύ. την κυρία Νάλεντι Παντόρ. Εδώ και ένα περίπου μήνα μια αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής επισκεφθήκαμε τη Ρουάντα και είδαμε τις πολιτικές που ακολουθούνται εκεί στον τομέα της ισότητας. Είχαμε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με μια πραγματικότητα. Είδαμε πώς οι γυναίκες μπορούν να γίνουν πρωταγωνίστρες της αλλαγής Επισκεφθήκαμε συγκεκριμένα κέντρα και πρωτοβουλίες, πήγαμε και σε ένα κέντρο κατάρτισης γυναικών και εκεί μια νέα είπε ότι το όνειρό μου είναι να είμαι μια ανεξάρτητη γυναίκα. Γι' αυτό ακριβώς η κατάρτιση και η εκπαίδευση είναι προϋπόθεση. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν στις γυναίκες τα μέσα έτσι ώστε να γίνουν μέσο για τη λύση των προβλημάτων μας στο μέλλον. Δεν ζητάμε πολλά, είναι νομίζω βασικός ο τομέας αυτός και εμείς που είμαστε υπεύθυνοι πολιτικά σε ορισμένα θέματα θα πρέπει να φωτίζουμε τις πρωτοβουλίες οι οποίες εντάσσονται στις αρμοδιότητές μας. Απαιτείται λοιπόν μια μεγάλη πορεία, μια δύσκολη πορεία και γι' αυτό απαιτούνται και μέσα και διευκολύνσεις για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας και θα περάσω τώρα στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Μάρια Μακάροφ μέλος του προγράμματος Norforsk που ασχολείται με την προβληματική των φύλων. Και μετά θα γίνει συζήτηση από τους συναδέλφους, θα πάρουν το λόγο εφόσον το επιθυμούν. Έχετε το λόγο. Μπορεί να έχω και διαφάνειες παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ας δούμε πρώτα τι είναι οι βόρειες χώρες. Είναι η Δανία στο νότο, Φιλανδία στη Δύση, Ισλανδία, ε, Φιλανδία στην Ανατολή, Ισλανδία στη Δύση, Σουηδία, Νορβηγία στο κέντρο. Τρεις από αυτές τις χώρες είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν όμως και αυτόνομες περιοχές. Ανάμεσα στη Σουηδία και τη Φιλανδία, μετά ε, τα νησιά όλων υπάρχει, υπάρχουν νηφερόες κάτω από την Ισλανδία και η Γρυλανδία στα βορειοδυτικά. Έχουμε 26 εκατομμύρια ε, κατοίκους και είμαστε από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίω. Οι βόρειες χώρες μοιράζονται πάρα πολλά κοινά στοιχεία πολιτισμικά, ιστορικά, ηθικές αξίες αλλά και έρευνα. Έρευνα που βασίζεται σε δημόσια παιδεία, σε δημόσια πανεπιστήμια. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φίλων στις βόρειες χώρες ε, ισχύει κάτι που δεν θα περίμενε κανείς. Οι βόρειες χώρες ε, είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη ισότητα στα δύο φύλλα στην Ευρώπη. Αν δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση, θα δούμε δείκτες οι οποίοι ε, δείχνουν ότι υπάρχει ισότητα. Αυτοί οι δείκτες ε, χρησιμοποιούνται και παγκοσμίως και όπως θα δείτε έχουμε πάνω από 70 στις βόρειες χώρες, ενώ οι υπόλοιπες χώρες ε, φτάνουν μέχρι το 60. Τώρα, ποιο είναι το παράδοξο. παρά το γεγονό ότι σε γενικέ γραμμές υπάρχει ισότητα των φύλων, δεν υπάρχει ισότητα στον πανεπιστημιακό χώρο. Περίπου η μισή απόφοιτη πανεπιστημίου είναι γυναίκες, ωστόσο οι ανώτερες βαθμίδες καθηγητών ανήκουν σε άνδρες τα ποσοστά εδώ πέφτουν από το 50% στο 24% συμμετοχής γυναικών σε ανώτατες καθηγητικές βαθμίδες, ενώ ε, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 20%. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η έλλειψη γυναικών σε καθηγητικές έδρες είναι μεγάλη. Δεν υπάρχουν πριτάνεις, δεν υπάρχουν ε, επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων. και δεν υπάρχουν γυναίκες που να καθορίζουν την επιστημονική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι οι πολύ σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο της ε, έρευνας και οι προτεραιότητες που καθορίζονται, καθώς και η χρηματοδότηση για αυτές, λαμβάνονται από το 50% της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, η πολυμορφία είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλους ε, τους τομείς και λήψη αποφάσεων και αν δεν υπάρχει ισότητα τότε χάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση. Τώρα, οι βόρειες χώρες προσπαθούν να επιλύσουν το ζήτημα αυτό της ε, ανισότητας, της μίσης εκπροσώπησης των φίλων στο πανεπιστημιακό χώρο. Μπορούμε να δούμε την εξής ε, προσέγγιση. Το 2013 το Ερευνητικό Συμβούλιο της Νορβηγίας σε συνεργασία με την Nordforsk, που θα σας εξηγήσω τι σημαίνει σε λίγο, δημοσίευσε μία έκθεση που περιείχε ανάλυση της ισότητας των φίλων στον ερευνητικό χώρο. Εδώ εντοπίστηκαν τρία κυρία σημεία. Η πρόοδος για την ισότητα των φύλων έχει ε, λιμνάσει και αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια. Έπειτα η ποιότητα της έρευνας που ε, διεξάγεται από γυναίκες έχει αλλάξει. Είναι εξίσου σημαντική με την πρόοδο της έρευνας των ανδρών, αλλά πολύ λιγότερη. Έπειτα, πολύ λιγότερες γυναίκες καταφέρνουν να ανελιχθούν στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης. Τώρα, τι κάνουμε εμείς, η Nordforsk, είμαστε ένας οργανισμός για διασυνοριακή ερευνητική συνεργασία στις βόρειες χώρες. Έχουμε μια πολιτική εντολή, διότι η Nordforsk βρίσκεται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Βόρειων Χωρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα, η Nordforsk έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί δύο κέντρα αριστείας για όλες τις βόρειες χώρες, δίδονται επιχορηγήσεις και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα που παρατηρείται στην ισότητα των φύλων. ασχολούμαστε με ανάλυση των συστημάτων καινοτομίας και έρευνας, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια και να καταλάβουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν για, για τα δύο φύλλα στην αγορά εργασίας και ε, τις ε, προκλήσεις που υπάρχουν στη χάραξη πολιτικής ισότητας. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε ότι η τρίτη κυρία δραστηριότητά μας αφορά το νομοθετικό έργο. Στη Φιλανδία από το 1995 η ισότητα των φύλων βρίσκεται αγκυροβολημένη στην νομοθεσία της χώρας. Η, για παράδειγμα, τα ερευνητικά συμβούλια τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση στην έρευνα πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον ε, κατά το 40% από ε, γυναίκες, από το υποεκπροσωπούμενο φύλλο. Έπειτα, η αιτήσει για ερευνητικά προγράμματα, ερευνητικέ επιχορηγήσει από τι γυναίκε έχει αυξηθεί. Τώρα το 50% των αιτήσεων γίνεται από γυναίκε, κάτι που δεν ίσχυε πριν τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, παρακολουθούμε τι εξελίξει και να ελέγχουμε τα ποσοστά ισότητας. Τώρα, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα προς ε, γυναίκες έχουν ως εξής. 50% συμμετοχή γυναικών σε μεταδιδακτορικά προγράμματα, περίπου 50% των επιτυχών αιτήσεων για αυτά τα προγράμματα είναι από γυναίκες, αλλά σε ό,τι αφορά τις ε, καθηγητικές έδρες, περίπου το 25% από αυτό είναι στελεχωμένο από γυναίκες. Εδώ παρατηρούμε δηλαδή ότι όσο πιο υψηλό το κύρος μιας θέσης, τόσο λιγότερες γυναίκες ε, κατέχουν τις θέσεις αυτές. Έπειτα, κοιτάζουμε την ίση εκπροσώπηση των δύο φίλων τα ανώτερα εκπαιδευτικά ειδήματα, στα ερευνητικά προγράμματα και βλέπουμε ότι και εδώ ισχύει αυτό το ε, περίεργο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βόρειων χωρών. Δηλαδή, όσο πιο ψηλέ οι θέσεις τόσο λιγότερη η εκπροσώπηση των γυναικών, παρά το γεγονός ότι η ισότητα είναι πολύ ε, μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, προσπαθούμε να εντάξουμε τη διάσταση του φίλου σε όλες τις ε, πολιτικές. Αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία η Σουηδία. Το 2015 μάλιστα ψηφίστηκε νόμος για την ίση συμμετοχή των γυναικών. Και είχαμε την πρώτη φεμινιστική, αν θέλετε, κυβέρνηση που έκανε πράξη αυτές τις συστάσεις για ισότητα των δύο φίλων. Αυτό διαφαίνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής και στον προϋπολογισμό. Αυτά όμως θα ε, σας ε, τα πούν αύριο οι συνάδελφοι από τη Σουηδία. Τώρα, η τελευταία μου διαφάνεια ε, παρουσιάζει μια πολύ σημαντική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή την έλλειψη των γυναικών στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, μηχανική. Οι γυναίκες και τα κορίτσια υποεκπροσωπούνται και στις σπουδές των θετικών επιστημών. Αυτό αρχίζει από το σχολείο. Οι γυναίκες λοιπόν λείπουν από μια αγορά εργασίας που εξελίσσεται ταχύτατα και αναπτύσσεται εξίσου ταχύτατα δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας στις θετικές επιστήμες κάθε χρόνο, νέες θέσεις εργασίας και σε ό,τι αφορά την ψηφιακή αγορά αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 800.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Και οι γυναίκες εάν δεν συμμετέχουν δεν σπουδάζουν σε θετικές επιστήμες δεν θα μπορούν να στελεχώσουν αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν συμπερασματικά θα μπορούσα να πω ότι χωρίς προορατικά μέτρα για την ισότητα θα πάει χαμένο το, το 50% του ταλέντου στις θετικές επιστήμες, στην καινοτομία, στις, ε, στους νέους τομείς δηλαδή που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την ευμερία. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Μακάροφ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι τα δεδομένα τα οποία μας καταθέσατε δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία θα πρέπει ε, να σταθούμε θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο οι γυναίκες και στην τεχνολογία και στην έρευνα. Ο αριθμός των γυναικών που ε, εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι ουσιαστικά χαμηλότερος των ανδρών. Μέσω λοιπόν του gender mainstreaming και εφόσον οι γυναίκες θέλουμε να συμμετέχουν στις διαδικασίες και στις αλυσίδες λήψης απόφασης θα πρέπει να ληφθούν ακόμα περισσότερο μέτρα. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στη συζήτηση θα σας δείξουμε ένα βίντεο. Ο Επίτροπος Μοέδας, ο υπεύθυνο Επίτροπος για την Καινοτομία και την Έρευνα θα μας στείλει το μήνυμά του. Δυστυχώς είναι, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις αλλού και γι' αυτό μας στέλνει αυτό το μήνυμα. We welcome the fact that the proportion of women in senior academic positions is steadily increasing. The number of women leading EU higher education institutions rose from 15% in 2010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 Bueno, pues una vez escuchado el mensaje del señor comisario, al que queremos agradecer, por supuesto, que haya querido trasladar. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω λοιπόν τον Επίτροπο για τα καλά του λόγια. Έχουμε γύρω στα 20 λεπτά για συζήτηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, για τη σημερινή διοργάνωση. Ήταν εξαιρετικές και οι δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε. Και οι δύο παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όπως έλεγα. Και από συναισθηματική ε, πλευρά ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Στην Ουγγαρία, στη χώρα μου, συχνά συναντώ ε, δυσαρεστημένες γυναίκες. Γιατί είναι δυσαρεστημένες, διότι δεν έχουν δουλειά ή γιατί δεν πληρώνονται αρκετά καλά. Και δεν αισθάνονται ασφάλεια και κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει τελικά. Οπότε, χρειαζόμαστε ακόμη πολύ περισσότερες προσπάθειες για να έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει ικανοποίηση και ικανοποιητικές αποδοχές. Πρόεδρε, η επιστήμη, η τεχνολογία, η καινοτομία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο τομέας όπου θα πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Να υπερβούμε αυτά τα προσκόμματα που ε, εμποδίζουν ε, την πρόσβαση για τις γυναίκες, είτε μιλάμε για την παιδεία, είτε για την αγορά εργασίας με άγγιξαν αυτά που είπατε και στις δύο παρουσιάσεις, ε, διότι και η δική μας η χώρα βιώνει βαθιές ε, πολιτικές ε, αλλαγές. Θα ήθελα να σας δείσω μια ειλικρινή απάντηση στο εξή ερώτημα. Μετά τις πολιτικές αλλαγές, πώς το βιώσατε. Είπατε εσείς, εμείς οι γυναίκες θέλουμε να προχωρήσουμε στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας και Δεν θέλουμε να εκμεταλλεύονται οι άλλοι ε, τις δεξιότητές μας. Δεν θέλουμε άλλοι να εκμεταλλεύονται τους ε, πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους. Θέλουμε εμείς να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους ε, και το εργατικό δυναμικό. Θέλουμε να πετύχουμε ε, ικανοποιητικές απολαβές ε, για τις νέες θέσεις εργασίας. Οι υποτιθέμενοι επενδυτές ε, έφεραν θέσεις εργασίας εξαιρετικά υποβαθμισμένες στην Ουγγαρία. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε άγουσα και να χαράξουμε μια πορεία προς την έρευνα, τεχνολογία και την καινοτομία Θέλουμε να ε, σχεδιάσουμε καινοτόμα προϊόντα, θέλουμε να τα θέσουμε σε εμπορία και να αποκομίσουμε τα ωφέλη από αυτή την προσπάθεια. Όταν αποφασίσετε να χαράξετε αυτή την πορεία στη δική σας χώρα, ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος των γυναικών, σας ρωτώ, διότι στην Ουγγαρία. Η επιστήμη και η οικονομία είναι συνειφασμένες με διαφθορά. Αυτό ε, το πρόβλημα πρέπει να υπερπηδήσουμε για να ακολουθήσουμε τον δρόμο της ε, ε, δικαιοσύνης και ισότητας στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας και της καινοτομίας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω περισσότερο από τις δικές σας εμπειρίες. η πρώτη φεμινιστική κυβέρνηση στον κόσμο. Αναφερθήκατε σε αυτό. Πρόεδρε, ε, πώς το επιτυγχάνει κάποιος αυτό, πώς επιτυγχάνει ε, κανείς ε, ικανοποιητική εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, ε, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε καλές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, ομιλίες σας. Πραγματικά εν, με ενέπνευσαν και στοχεύουν να φέρουν περισσότερες γυναίκες στον χώρο της επιστήμης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε στην Ευρώπη να επιτύχουμε και ελπίζω η ε, καλή διάθεση που έχουμε δείξει να συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε πολύ περισσότερες γυναίκες να μπουν στον χώρο των επιστημών, στον χώρο της ε, λήψης αποφάσεων, σε αυτό το χώρο στις θετικές επιστήμες. Ε, και μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι παρά το γεγονό ότι οι Σκανδιναβικέ, οι βόρειε χώρε ε, ε, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ισότητα, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στι ηγητικές ε, θέσεις που οι γυναίκε υποεκπροσωπούνται. Αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολο και σοβαρό είναι το ναι. πρόβλημα. Πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες, διότι έτσι θα αλλάξει η κοινωνία, θα υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία. Και πιστεύω πως εδώ το πρόβλημα είναι ότι ίσως μας λείπει όχι η θέληση αλλά τα μέτρα. Τα μέτρα δηλαδή που θα γίνουν νομοθεσία και θα οδηγήσουν στην ε, ισότητα. Υπάρχουν, ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα που θα μας ε, πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιος άλλος το λόγο. Εσείς, συγχωρέστε με που δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα, αλλά ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνα της Ιταλίας θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η Σνάουντερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει μια εξαίρετη προσπάθεια έχει βοηθήσει να τις χώρες έτσι ώστε να λειτουργήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις υποδεγματικά. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο θα γίνονται οι παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να κάνουν ε, τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά θα πρέπει και τα δημόσια όργανα να παίρνουν πρωτοβουλίες. Πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες να προωθήσουν σαν παράδειγμα το Gender Equality Plan. Το θέμα είναι θέμα πολιτισμικό, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα αντίληψης και αυτού του είδους τα προβλήματα δύσκολα αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά και γρήγορα. Ίσως και θα χρησιμοποιήσω ένα ρήμα όχι πολύ δημοφιλές. Πώς θα υποχρεώσουμε, πώς θα εξαναγκάσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε όλες αυτές οι δραστηριότητες να ενσωματωθούν στην λειτουργία των κρατικών οργάνων, των δημοσίων οργάνων. Ευχαριστώ τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Είμαι από το Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας. Ασχολούμαι με το θέμα, κάνω έρευνα για το θέμα της θέσης των γυναικών στις ερευνητικές διαδικασίες, στις ερευνητικές δραστηριότητες. Οι έρευνες μέχρι τώρα μας δείχνουν ότι σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις έρευνες μας. Στοιχεία τα οποία δείχνουν επίσης ότι μπορεί ε, εφόσον βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών να βελτιωθεί και η παραγωγικότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας Υπάρχει εδώ ένα θέμα που συνδέεται, είναι η νοοτροπία, η πρακτική η οποία ακολουθείται για υπερβολικά πολύ μεγάλα ωράρια εργασίας. Πέφτουν θύματα οι γυναίκες αυτής της πρακτικής. και επηρεάζει αρνητικά την ε, οικονομική δραστηριότητα και τοπικά και γενικότερα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε λοιπόν, να στοχεύσουμε σωστά το συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί με τέτοιου είδους αντιλήψεις, ε, οικονομικές δραστηριότητες ε, και τέτοιου είδους μορφές επιδιωκόμενης αποδοτικότητας ε, δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω θέσεις για τις γυναίκες στον τομέα της έρευνας. Επίσης ε, σε επίπεδο χρηματοδότησης θα πρέπει οι ανθρωπιστικές επιστήμες να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο γιατί έμεσα αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν είναι τόσο πρακτικά όσο κοινωνικά. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτού του είδους τις επιστημονικές σπουδέ να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θα συμφωνήσω πλήρως με την τελευταία παρέμβαση και η υπουργό εδώ δίπλα μίλησε για τον προσωρινό χαρακτήρα όχι μόνο της απασχόλησης σε γενικό επίπεδο αλλά και στον τομέα της έρευνας. Αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στα πλαίσια μιας έκθεσής μας πρόσφατα η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης, η πολιτική της λιτότητας, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές βλάβες σε ορισμένους τομείς, είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό εμείς μιλάμε για τομείς της κοινωνίας, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και η πολιτική αυτή των περικοπών ουσιαστικά δεν βοηθάει καθόλου. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε σε μια νέα πολιτική αντίληψη που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της επενδυτικές και να καταπολεμήσουμε τον προσωρινό χαρακτήρα των μέτρων που λαμβάνουμε στα πλαίσια των εργοσιακών ρυθμίσεων. Γιατί όπως είπα δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες είναι απολύτως άδικες και αδικαιολόγητες. Τώρα θα δώσω το λόγο στις ε, ομιλήτριες, προς τις οποίες απευθύνθηκαν ορισμένες ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσουν γρήγορα να απαντήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθησαν. Σίγουρα η οικογένεια έχει πρωταρχική σημασία, αλλά να πω πως είδα τα βιογραφικά ορισμένων πραγματικά ιδιοφυλιών των μαθηματικών που έζησαν στην Ευρώπη τα τελευταία 100 χρόνια. Και ξέρετε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό τους, ότι είχαν γονείς πατέρα που τους στήριξε. Και αυτό έγινε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται πως οι υποδομές είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση. Αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να ε, εξετάσουν οι υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής. Τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πέρα από τη Σουδία και τη Φιλανδία η Νορβηγία πριν από κάποια χρόνια ψήφισε ποσοστώσεις για τον ιδιωτικό τομέα, για, ε, την εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Ψήφισε λοιπόν μια ποσόστοση 40% εκπροσώπησης τουλάχιστον από γυναίκες. Τώρα, αναφέρθηκαν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ναι, σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε. Η ηγεσία των ε, θεσμικών οργάνων πρέπει να ασχοληθεί με αυτή την προβληματική, το πώς δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί μια οικογένεια με παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία. Τώρα, ε, να επανέλθω στα χαμηλά ποσοστά των συμμετοχή ε, συμμετοχής γυναικών στα κέντρα αριστείας των βορείων χωρών. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της έρευνας, ε, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν να υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες εφόσον η ποιότητα της έρευνας είναι εφάμιλοι με εκείνη των ανδρών. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες και να δούμε πολλά κριτήρια. Ε, να δούμε για παράδειγμα ε, άλλους τομείς όπου ε, παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση. Πιστεύω πως το θέμα είναι πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Στη Φιλανδία, τη χώρα μου, η συμπεριφορά των ερευνητικών συμβουλίων που είναι ο κύριος φορέας ε, ενίσχυσης των ερευνών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, όταν γίνεται μία αίτηση για ερευνητικό πρόγραμμα θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να στηρίζει την ισότητα, να υπάρχει ένα σχέδιο που να εφαρμόζεται πολιετές. και να διασφαλίζεται ότι θα εφαρμόζονται αυτές οι προδιαγραφές ισότητας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενσωματωθεί μέσω της νομοθεσίας η ισότητα στο ε, σύστημα. Έτσι μπορούμε, πιστεύω, να συνεισφέρουμε στην ε, αλλαγή των ποσοστών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, μία ερώτηση είχε τεθεί σε μένα για την καινοτομία και το αν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια καινοτόμως οικονομία όπου θα υπάρχει προστιθέμενη αξία πέρα από τους φυσικούς πόρους και τα αγαθά που μπορεί να παραγεί η χώρα μας. Είναι μια πρόκληση για την Νότια Αφρική, διότι είμαστε περισσότερο προσανατολισμένοι στα αγαθά και από τη στιγμή που τελειώσει ο χρυσός ή η πλατίνα τότε η χώρα μας θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Θα ε, αλλάξουν τα δεδομένα, θα αυξηθούν οι τιμές, αυτό το έχουμε δει σε άλλες χώρες της Αφρικής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε ικανότητα να ε, η καινοτομία να επιφέρει προστιθέμενη αξία. Προσπαθούμε λοιπόν όχι μόνο να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία της ε, καινοτομής αυτής, αλλά και να αλλάξουμε την ε, οικονομία μας. Αυτή τη στιγμή στη Νότια Αφρική η πλατίνα είναι ένας φυσικός πόρος σε αυθονία και προσπαθούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην τεχνολογία, ιδιαίτερα σε ε, κυψέλες ε, ενεργειακές. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται η πλατίνα σε αυτές τις ε, ενεργειακές κυψέλες που θα αντικαταστήσουν τους υδρογονάνθρακες. Αυτό πιστεύουμε θα επιφέρει προς τη θέμενη αξία στην νέα εκβιομηχάνηση της ε, οικονομίας της Νοτιοφρικής και στον μεταποιητικό τομέα. Φυσικά χρειάζεται και να δούμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Νοτιοαφρική θα θέλαμε να αυξηθούν οι εξαγωγές, όμως πρέπει να, ε, να γνωρίσουμε πώς χρειάζονται και οι εισαγωγές. Δεν είμαστε απομονωμένη χώρα και σίγουρα θα ήταν απατηλό να πιστεύαμε πως η οικονομία μας μπορεί να ε, στηριχτεί και να εξελιχθεί αυτόνομα. Γι' αυτό λοιπόν είναι φανερό πως χρειάζεται η έρευνα για να στηριχθεί η οικονομία. Χρειάζεται έρευνα, αλλά πρέπει επίσης και να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στον ε, υπόλοιπο κόσμο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μας λοιπόν στην Νότια Αφρική χρησιμοποιήσαμε το εξή απόφθεγμα. Πρέπει να προχωράς αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς να υποχωρείς. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε πώς ε, για να προχωρήσουμε πολλές φορές χρειάζεται να υποχωρήσουμε είναι τώρα πολύ σημαντικό να δούμε τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μα ή που μπορούμε να λάβουμε και να διασφαλίσουμε ότι ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικό. Αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των κοινοβουλίων και θα έπρεπε να ε, το έχουν υπόψη αυτό. Τα κοινοβούλια εκλέγονται από το λαό με την εντολή να ασκούν έλεγχο και να χαράσουν πολιτική. Η πολιτική όμως δεν είναι δράση. Η πολιτική εμείς δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε οι πολιτικές που δημιουργούμε να έχουν θετικές επιπτώσεις στο, στον κόσμο, στον πληθυσμό. Έχουμε τελειοποιήσει τη χάραξη πολιτικής, δυστυχώς όμως έχουμε τρομερές ελλείψεις στην υλοποίησή της και τον έλεγχο. Χρειάζεται λοιπόν οι πολιτικές που χαράσουμε να φροντίζουμε να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία, να αλλάξουν τις ζωές των γυναικών, να εφαρμοστούν στην πράξη. Αυτό είναι έργο όλων και καθήκον όλων των κοινοβουλίων σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. τα τελικά συμπεράσματα του πάνελ θα δώσω το λόγο στον κύριο Πίντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Συζητήθηκε το θέμα της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί και των αλλαγών στην πολιτική. Απαιτείται να υπάρξουν ριζικές δράσεις για να πετύχουμε τις αλλαγές Τέθηκε το θέμα των επίσημων δεσμευτικών προγραμμάτων και σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να τα σεβαστεί και να τα εφαρμόσει πλήρως. Έχουμε κάποια παραδείγματα και στον Καναδά, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, έτσι ώστε τα όργανα να έχουν τέτοιου είδους προγράμματα ισότητας κατά τη λειτουργία τους αν και να υπάρχουν και συνέπειες, να υπάρχουν κυρώσεις στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνονται σεβαστά και πώς θα πρέπει οι πολιτικές αυτές να εφαρμόζονται. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ριζικές παρεμβάσεις και οι πολιτικές παρεμβάσεις είναι από τα πιο χρήσιμα μέσα στον Καναδά. Οι 15 από τους 31 υπουργούς στον Καναδά είναι γυναίκες τώρα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Υπάρχει και ένα ειδικό υπουργείο που ασχολείται, η κυρία Πετρούσα Χάτζη είναι υπουργό γυναικείων θεμάτων. Η υπουργό έρευνα, η κυρία Ντάνκαν, είπε πριν τρει εβδομάδε ότι θα ακολουθήσουν δεσμευτικέ πολιτικέ ρυθμίσει έτσι ώστε ε, όταν είναι να ανοίξουν νέου τύπου ε, υψηλού επίπεδου ερευνητικές θέσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από προγράμματα ισότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή Υπάρχει μια αιμονή με την παραγωγικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε και γι' αυτό. Σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε αν θέλετε τους συναδέλφους στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών, στα πλαίσια των προκαταλήψεων συνειδητών ημί και θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών σταδιοδρομιών και δεν θα πρέπει να είμαστε αιμονικοί με την παραγωγικότητα και νομίζω ότι συλλογικά και συνεργατικά θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Ήταν μεγάλη χαρά λοιπόν που παρακολούθησα τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να κηρύξω την λήξη των εργασιών αυτού του πάνελ. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμμετοχή σας εδώ. Ε, διακόπτουμε για ένα-δύο λεπτά για να υπάρξει εναλλαγή των προσώπων στο πάνελ.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

Vamos a comenzar esta sesión. No, se oye bien, ¿eh? Sí, los dos. Buenos días. Eh, vamos a comenzar este segundo panel, si Παρακαλώ καθίστε για το δεύτερο πάνελ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε εντυπωσιακέ παρεμβάσεις που θα κάνουν τις ε, ομιλίες για τις διαφορές ε, στον τομέα της υγείας ανάμεσα στα φύλλα. Συμπρόεδρος λοιπόν είναι η κυρία Νταμόνσε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, παρακαλώ, οι ιδιωτικές σας συζητήσεις εκτός εθούσης, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνει η Πρόεδρο στα αγγλικά, αν θέλετε να κάνετε ιδιωτικές παρεμβάσεις, να βγείτε εκτός εθούσης. Για μια ακόμη φορά λοιπόν σας καλωσορίζω. Όταν μιλάμε για έλλειψη ισότητας, μιλάμε συνήθως για διαφορές ε, ε, μισθοδοσίας, ε, αλλά υπάρχει και το θέμα της βίας, υπάρχει το θέμα της ψυχολογικής βίας, υπάρχει και το θέμα της υγείας. Υπάρχουν λοιπόν στον συγκεκριμένο τομέα διαφορές ανάμεσα στις άνδρες και τις γυναίκες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η υγεία είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής, οικονομικής και σωματικής ευημερίας. Ε, υπάρχουν διαφορές και σε θέματα γενικότερα αναπηρίας, αλλά θα μιλήσουμε για το κύριο θέμα, το οποίο είναι το θέμα της υγείας. Υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα πολλές φορές ε, στον τομέα της υγείας. Το θέμα της ενδομητρίωσης, ας πούμε, είναι αποκλειστικά γενικείο και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την συγκεκριμένη πάθηση. Τίθενται λοιπόν ε, ε, αντίστοιχα προβλήματα και για άλλες ασθένειες και βλέπουμε ότι υπάρχουν διακρίσεις γιατί η ανδρική ανικανότητα σαν παράδειγμα συγκεντρώνει πολύ περισσότερες πιστώσεις διαρευνητικές από ότι η ασθένεια της ε, ενδομητρίωσης της γυναίκες. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει έλλειψη γενικά στον τομέα της υγείας των απαραίτητων υποδομών. Αυτό λειτουργεί εις βάρος των γυναικών. και στα πλαίσια της αναπαραγωγικής υγείας δημιουργούνται πολύ σημαντικά θέματα σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περικοπές στο σύστημα πρόνοιας έχει χτυπήσει την γυναίκες και έχει χειροτερεύσει την κατάστασή τους. Είναι σαφείς λοιπόν οι διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες αναφερόμαστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίμιση δηλαδή του πληθυσμού και ενώ υπάρχουν θεωρητικά δικαιώματα αντίστοιχα και ισότιμα σε όλους τους τομείς, στον τομέα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων ε, τα πράγματα είναι σε διαφορετική κατάσταση και ο ρόλος των γυναικών σε υψηλές θέσεις ευθύνης είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τους άνδρες πόσες γυναίκες είναι υπεύθυνε για μεγάλα νοσοκομεία ή για μεγάλες φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Γενικότερα λοιπόν ε, υπάρχουν βέβαια και ορισμένες καταστάσεις αντίστοιχες όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες σε σχέση με την ε, κατάθλιψη ή σε σχέση με τις συνέπειες της προκεχωρημένης ηλικίας αλλά παρόλα αυτά οι διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο παραμένουν σημαντικές. Ε, οι γυναίκες οι οποίες ζουν σε ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον θα έχουν στη συνέχεια και, μια, και περισσότερες πιθανότητες για μια κανονική ψυχολογική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να κάνει τα απαραίτητα, θα πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες μέλη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των αναπηριών και να προωθήσει την σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των γυναικών όταν καθορίζονται τα πολιτικά μέτρα στον τομέα της υγείας. Αυτό είναι μια ευθύνη και πολιτική και κοινωνική σε όλα επαναλαμβάνω τα επίπεδα και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εθνικό ή Έχουμε τις δυνατότητες να παρέμβουμε και να βρούμε λύσεις. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικό σύνολο ομιλητών. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο όμως στην κυρία Ντεμονσέ, η οποία με συνοδεύει. Είναι τιμή μου που συμπροεδρεύομαι σήμερα. Είναι Group Executive του Science Engagement του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας της Νοτιού Αφρικής. Εδώ και 10 χρόνια υπηρετεί στην συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι μέλος επίσης του Φόρουμ Γυναικών της Νοτιού Αφρικής, του Συμβουλίου Επιστημών της Νοτιού Αφρικής. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Νταμόνσε. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Μπέβερλι, έχεις το λόγο, μπορείς να κάνεις και εσύ μια εισαγωγή ως συμπρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και ευχαριστώ και τη Σύνοδο για τη σημερινή διοργάνωση. Ε, 20 χρόνια τώρα έχουμε ολοκληρώσει το πέρασμα στη συνταγματική δημοκρατία από το ότι Αξιοσημείωτη κοινωνική πρόοδο έχει γίνει για την ανατροπή όλων αυτών των πρακτικών που διεύθυνουν κάθε πτυχή τη κοινωνική ζωή και υποβάθμιζαν το ευσύν όλων των Νότιο-Αφρικανών και θα πρέπει να υποτιμούμε ε, το βάρος των ε, μεταδοτικών ασθενειών που είναι αντίθετες ε, προς αυτό το μοντέλο που θέλουμε να επιτύχουμε στον τομέα της υγείας. Ε, πώς πρέπει λοιπόν να κινηθούμε και ποιες είναι ποιε είναι οι άμεσε και έμεσε σχέσει ανάμεσα στην υγεία και την κοινωνική ευημερία. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκε αυτέ οι σχέσει. Όταν η ακραία φτώχεια πλήττει ε, τα κοινωνικά στρώματα, τότε υπάρχει έλλειψη πρόσβαση σε βασικές απαιτήσει, σε καθαρό πόσιμο νερό, κατάλληλη ε, σύντηση, αποχετεύσεις, ε, κατάλληλα καταλήματα, εμβολιασμό, καλά σχολεία και όλα αυτά μας οδηγούν στη μη διαθεσιμότητα καλών θέσεων εργασίας και μείωση του προσδοκίμου ζωής. Ε, βλέπουμε ότι η υγεία λοιπόν συνδέεται άρρηκτα με τον κοινωνικό ιστό και με τις δυνατότητες που αναπτύσσουν ή ένα έθνος χάρη στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Νομίζω ένα από τα βασικότερα άχθη που φέρουμε είναι οι ανισότητες που γνωρίζει η χώρα μας ε, κυρίως για νοσήματα όπως το AIDS. 0,7% ε, του παγκοσμίου πληθυσμού, τουλάχιστον όμως 17% των κρουσμάτων ε, AIDS. Στο κέντρο της ε, ε, επιδημίας είναι οι έφηβες ε, και νέες γυναίκες 15 ή 24 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι ανισότητες αποτυπώνονται και στις τάσεις της πανδημίας αυτής αυτή ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των κοριτσιών και νέων γυναικών ε, περνούν από πάρα πολύ δύσκολες φάσεις ορίμανσης ε, ε, και είναι ιδιαίτερα ευπαθείς αυτές οι γυναίκες σε αυτή την μεταβατική περίοδο. Λοιπόν, για τις τάσεις ως προς την αρρώστια αυτή, νομίζω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ε, ε, αντιστοιχούν στο 42% των, ε, της θνησιμότητας ε, των μητέρων ε, και γιατί έχουμε και τη μετάδοση στα έμβρια και φυσικά έχει επιτυχθεί η μείωση του 2% όμως διαπιστώνουμε ότι οι μεταδοτικές ασθένειες ε, είναι ένας ε, τομέας όπου κατεξοχήν θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και την υγεία αυτών των κοριτσιών και νερών γυναικών, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για το καλό της χώρας μας. Muchísimas Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νταμόνσε. Θα δώσω τώρα το λόγο στις προσκεκλημένες μας, κυρία Ρόμπι Νόρτον, του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Υγεία, μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σαν στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης πρόνοιας και συνδρομής. είναι στα δέκα πιο γνωστά Ινστιτούτα τα οποία έχουν αξιολογηθεί στον συγκεκριμένο τομέα στον κόσμο. Μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μποτρούβα, υπεύθυνη της συγκεκριμένη πρωτοβουλία SPG από το Λονδίνο. Είναι επίσης και σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών για την εξέταση και μεγαλύτερη λήψη υπόψη των θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Νόρτον μέχρι 15 λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Νόρτον δεν ακούγεται. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο οργανωτές για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι χαρά μου που ε, είμαι μαζί σας. Θα ήθελα να αρχίσω με μια διαφάνεια και να σας πω πρώτα πως έχω δύο μηνύματα να δώσω στο ακροατήριο σήμερα. Πρώτον, ότι τα κύρια αίτια θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες παγκοσμίω Τώρα είναι νοσήματα ε, μη μεταδιδόμενα. Έπειτα, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτό το πρόβλημα των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων που αποτελούν αιτία θανάτου για τις γυναίκες, πρέπει να δούμε ε, την διάσταση του φύλου στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με την υγεία, έτσι ώστε να βρούμε τρόπο να αποτρέψουμε αποτελεσματικά ε, τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους ε, συντάκτες της έκθεσης μια έκθεση για την παγκόσμια υγεία που δημοσιεύτηκε ε, υπό την αιγίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου στις αρχές του έτους. Θα είναι αύριο εδώ στο πάνελ για να σας παρουσιάσουν την έκθεση αυτή. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια θα ήθελα να εστιάσω λίγο στα κύρια αίτια θανάτου για τις γυναίκες και κυρίως να σας μιλήσω για τα κύρια αίτια θανάτου για τις γυναίκες χωρίς να αναφερθώ στα αίτια θανάτου για τους άντρες. Και αυτό γιατί τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές που αντικατοπτρίζουν και τις ε, αλλαγές στην υγεία, στα συστήματα υγείας. Με επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό πόρων έχει διοχετευτεί στην μείωση της ε, θνησιμότητας των ε, γυναικών κατά τη γέννα. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές προσπάθειες για να μειωθεί και η θνησιμότητα των νεών και η θνησιμότητα της ε, μητέρας. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών και μειώθηκαν λοιπόν οι θάνατοι αυτοί κατά 45% από το 1990 μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια τεράστια αλλαγή ε, που βελτιώνει τη ζωή των γυναικών. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι ένα από τα κυριότερα αίτια θανάτου για γυναίκες δεν είναι κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα. Εφτά από, τις, ε, από τα 10 ε, κυριότερα αίτια θανάτου είναι μη μεταδιδόμενα νοσήματα ε, και τα κυριότερα αίτια θανάτου είναι διάφορες καρδιακές παθήσεις ή εγκεφαλικό. Υπάρχουν ε, επίσης αναπνευστικά προβλήματα τα οποία αποτελούν και αυτά ένα αίτιο θνησιμότητας. Επίσης, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να μειωθεί ο καρκίνος του μαστού Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τώρα ε, η κυριότερη, η μορφή καρκίνου που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Επίσης, η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η πέμπτη ε, μεγαλύτερη αιτία θανάτου για τις ε, γυναίκες. Τώρα, θα ήθελα να δώσω λίγο έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ιδιαιτερότητες της χώρας αυτής. Είναι μια χώρα πύκνο κατοικημένη και βλέπουμε ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο 9 στις 9 ε, στα 10 ε, αίτια θανάτου είναι μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο καρκίνος είναι είναι στην τέταρτη θέση και ο καρκίνος των πνευμόνων ε, η κυριότερη μορφή καρκίνου. Τρεις στους δέκα θανάτους επίσης οφείλονται στην νόσο του Αλτσχάιμερ, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη θανατηφόρος ασθένεια. Μετά, ας δούμε όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Ας δούμε τι συμβαίνει και στις χώρες με μεσαίο ή μικρό εισόδημα. Εδώ βλέπουμε πως τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα αποτελούν το 50% το οφείλ, το, αποτελούν το 50% των θανάτων. Τα μεταδιδόμενα όμως νοσήματα στις χώρες με μεσαίο και χαμηλό εισόδημα ευθύνονται για το υπόλοιπο 50% των θανάτων. Τώρα, θέλω να δώσω περισσότερη έμφαση στην Ινδία στην επόμενη διαφάνεια. Η Ινδία θεωρείται χώρα μεσαίου εισοδήματος παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, στην επικράτεια της χώρας, μισθολογικές. Εδώ βλέπουμε πάλι ε, πως ε, οι καρδιοπάθειες και τα κεφαλικά είναι οι ασθένειες με τους περισσότερους θανάτους. Αναπνευστικές παθήσεις επίσης, 4 στους 10 θανάτους στην Ινδία. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα θα έπρεπε να είναι στην ε, κορυφή των προτεραιοτήτων μας εάν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ε, υγεία των γυναικών. θα περίμενε κανεί πω και οι κυβερνήσει και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι ίδιε οι γυναίκε θα ε, ζητούσαν οι ίδιες να γίνει κάποια αλλαγή στην κατάσταση και να είναι καλύτερα ενημερωμένε. Βλέπουμε όμως ότι και από τη μία και οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέτουν ως προτεραιότητα την μείωση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και αντίστοιχα η πολιτική. Επίσης, θα περίμενε κανείς ότι η στρατηγική για τις ε, νέες ε, γυναίκες θα ανέφερε τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν κάποια ε, σημεία εστίασης για την υγεία των εφήβων, των παιδιών και των νέων, που πράγματι αφορούν τη μείωση των ε, μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και την βελτίωση της ψυχικής υγείας των γυναικών. Όμως υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι συνεχίζουν να επιμένουν ε, στην αναπαραγωγική υγεία, σεξουαλική υγεία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά πρέπει να βρούμε μία ισορροπία και ε, να συμπεριληφθούν και τα υπόλοιπα αίτια θανάτου για γυναίκες. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα είναι εξίσου ε, σημαντικά και εξίσου επιβλαβή για την υγεία τους. Έγινε μία έρευνα μάλιστα ε, κατά την οποία ερωτήθηκαν εάν οι διάφορες ε, νόση του κυκλοφοριακού συστήματος πλήττουν περισσότερο άνδρες ή γυναίκες. Οι απαντήσεις ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες, ανησυχητικές. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες καταλαβαίνουν πως οι διάφορες, ε, αυτά τα νοσήματα του κυκλοφοριακού συστήματος είναι πολύ σημαντικά. Από την άλλη όμως βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις άλλες χώρες με υψηλό εισόδημα υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι φτωχότεροι πάσχουν από εξίσου ε, από τις ίδιες ασθένειες με ε, εκείνες ε, που πλήττουν άλλες χώρες με χαμηλό ή εισόδημα. Τώρα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν επίγνωση του πόσο σημαντικές είναι οι καρδιαγκιακές παθήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά μα, να προσπαθήσουμε δηλαδή να εντοπίσουμε και να μεταδώσουμε στο κοινό το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ασθένειες και πόσο σημαντική, ακόμα σημαντικότερη, είναι η πρόληψη των ασθενειών αυτών. Και πραγματικά, όπως θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια, εάν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στα ε, δεδομένα που έχουμε για την υγεία. Τα δεδομένα αυτά και τα στατιστικά στοιχεία προς το παρόν αφορούν ως επιτοπλίστων άνδρες. Αυτό όχι μόνο αποτελεί ε, διάκριση, αλλά οδηγεί και σε ε, δυσάρεστες επιπτώσεις για την υγεία των γυναικών. Επόμενη διαφάνεια. Τι εννοούμε όμως με μία ε, διαφορετική προσέγγιση ε, που θα στηρίζεται στην ισότητα των φύλων ε, για την υγεία. Καταρχάς, υπάρχουν αναλύσεις που γίνονται κατά φύλο. Αυτές οι αναλύσεις και αυτές οι μελέτες μας έχουν βοηθήσει να εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Αυτές λοιπόν οι ξεχωριστές αναλύσεις μας έχουν ε, δείξει πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε άντρες και γυναίκες, οι οποίες διαφορές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες εκτός από τους ε, βιολογικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς κτλ. Έπειτα, η προσέγγιση αυτή που υιοθετήσαμε επικεντρώθηκε κυρίως ε, στις καρδιοπάθειες. Και είδαμε εδώ ότι ε, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άντρες για να πάθουν εγκεφαλικό σε μεγαλύτερες ηλικίε. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ως προς την ε, υγεία και ως προς τους ε, κινδύνους. Οι γυναίκες επίσης δεν παραπέμπονται τόσο συχνά όσο οι άνδρες σε διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Οι γυναίκες επίσης επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους άνδρες, ε, από τον ε, διαβήτη και από, το, και από τις συνέπειες του καπνίσματος. Και όπως θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια, ίσως δεν μπορείτε να δείτε ε, τα νούμερα γιατί είναι μικρά τα γράμματα, όμως βλέπουμε ότι οι γυναίκες διατρέχουν πρόσθετους κινδύνους από τα εμφράγματα, από το κεφαλικό, από τον διαβήτη τύπου 1 και 2 από ότι άντρε. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι γυναίκες που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 έχουν 40% μεγαλύτερο κίνδυνο για να πάθουν κεφαλικό από ότι άντρες με διαβίτη τύπου 2. Ας δούμε τώρα τη μελέτη που εστίασε στις ε, καρδιοπάθειες καρδιακές παθήσεις. Βλέπουμε αυτές τις διαφορές. Δεν περιμένω να διαβάσετε τις λεπτομέρειες αυτό το πίνακα, αλλά βλέπουμε σαν παράδειγμα ότι όταν βλέπει κανείς ε, τις ε, γυναίκες και τους άνδρες με διαβήτη, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ε, πρόβλημα και μεγαλύτερο κίνδυνο να πάσχουν από από σοβαρές ψυχικές ασθένειες από ότι οι άνδρες. Θα πρέπει να ελέγξουμε ακόμα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, να δούμε αν οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με τον ίδιο τρόπο με τους άνδρες. Μπορώ να έχω και την επόμενη διαφάνεια. Θα τελειώσω εδώ λέγοντας ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα θέματα αυτά να αρχίσουμε να τα συζητάμε όλο και περισσότερο και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υψηλού, υψηλών εισοδημάτων. Στην Ινδία τώρα ξεκινάμε να ελέγχουμε τέτοιου είδους βάσεις δεδομένων από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες για να δούμε ακριβώς τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις, στους άνδρες και τις γυναίκες. Ελπίζω μέσα στο λίγο χρόνο που είχα στην διάθεσή μου να σας έδειξα ότι οι βασικές αιτίες θανάτου και αναπηριών για τις γυναίκες και στις χώρες των μέσων εισοδημάτων και η ε, μη μεταδιδόμενες ασθένειες είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να κατανοήσουμε και να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας παρουσίαση όχι μόνο γιατί δεν ξεπεράσατε τον χρόνο τον οποίο είχατε στη διάθεσή μας, αλλά νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε το μέγεθος των προβλημάτων που έχουμε. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, δεν γνωρίζουμε το τι δεν γνωρίζουμε και ελπίζω ότι οι σκέψεις τις οποίες εκφράσατε και εσείς και τις οποίες εκφράζουμε και εμείς θα τα μεταφέρουμε και σε σχέση με τις ευθύνες τις οποίες έχουμε ε, εκτός αυτής της αιθούσης. Πολλές φορές τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ε, αν δεν είναι λανθασμένα, είναι μη χρηστικά και πολλές φορές ε, είναι μέτρα τα οποία αντικατοπτρίζουν διακρίσεις και δημιουργούν προβλήματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για το ίμιση του πληθυσμού των χωρών μας. Είναι δυστυχώς λανθασμένες ε, πολλές από τις πληροφορίες αυτές και όταν εργαζόμαστε με βάση λανθασμένα στοιχεία είναι προφανές ότι και τα αποτελέσματά μας δεν θα είναι ικανοποιητικά και αυτό θα βλάψει ακόμα περαιτέρω την υγεία των γυναικών. Νομίζω λοιπόν ότι το σημαντικό μήνυμα εδώ είναι η ποιότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε και γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες ε, που φροντίζουν για τις γυναίκες να γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να προσπαθήσουν να δουν ποια είναι τα προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία τους. Θα δώσω τώρα αμέσως το λόγο στην κυρία Μπότροβα μέχρι 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλημέρα. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της Συνόδου για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Τα ζητήματα ε, των δύο φίλων ε, μου ήταν ιδιαίτερα προσφυλή ανέκαθεν και χαίρομαι και είναι τιμή για μένα που μιλώ για την ε, ψυχική υγεία σε αυτή τη σύνοδο. Η Καμπριέλα θα προβάλλει τις διαφάνειες ε, για μας. Ε, ε, θέλω να κάνω δυναμικές παρουσιάσεις και θα δίνω τις εντολές για να προχωράει με τις διαφάνειες. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί σε μια τέτοια σύνοδο έχει σημασία η ψυχική υγεία. Όταν παρουσιάζω την, την ομιλία μου, ξύπνησα ε, το Σάββατο και κοιτάζω το λογαριασμό Twitter και βλέπω αυτό. Ε, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες, έλεγε στον Guardian, ε, για τους άντρες ε, να αναζητήσουν βοήθεια για την ψυχική υγεία από ότι οι γυναίκες. Αυτό είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας και επηρεάζει τους ανθρώπους. Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από τέτοιες ψυχικές διαταραχές. Θα ήθελα να διερευνήσουμε τις σχέσεις με τα ε, ζητήματα των φύλων, τη σχέση των ε, βιώσιμων στόχων της χιλιετίας ε, του ΟΗΕ και κυρίως σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους και επίσης να δούμε και τους δείκτες αυτών των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Γιατί είναι σημαντική η ψυχική υγεία. Πέντε λόγους θα σας δώσω. Είναι καταπήγον το ζήτημα. Ένα στου τέσσερις ανθρώπους υποφέρει κατά τη διάρκεια του από μια τέτοια πάθηση. 600 εκατομμύρια δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Η κατάθλιψη θα αναδειχθεί ε, μέχρι το 2020 στη δεύτερη σοβαρότερη ασθένεια. Επίσης, είναι θανατηφόρα τα νοσήματα. Υπάρχει ε, εξαιρετικά υψηλή θνησιμότητα. Για τους άντρες ε, πεθαίνουν 20 χρόνια νωρίτερα και οι γυναίκες 15 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με υγιείς ανθρώπους. Από χώρες υψηλού εισοδήματος έχουμε συλλέξει τα στατιστικά στοιχεία και κατά πάσα πιθανότητα από ε, χώρες χαμηλού εισοδήματος θα είναι πολύ χειρότερα τα στοιχεία και επίσης είναι η δεύτερη αιτία για αυτοκτονίες σε ηλικιακή κατηγορία 15 έως 29. Ας πάρουμε τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από τέτοια νοσήματα ζουν σε τέτοιες χώρες και 76-85% αυτών των ανθρώπων δεν, έχουν, ε, δεν ε, λαμβάνουν καμία αγωγή. Επίση, ε, κατάφορε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση, κοινωνική αποξένωση, αποκλεισμό, και βίες πρακτικές ε, όπως ε, παραδείγματος χάρη τους αλυσοδένουν στην Ινδία όπως βλέπετε σε αυτή την φωτογραφία. Επίσης ε, είναι εγκάρσιο το ζήτημα σε σχέση με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και έχει στενές σχέσεις με τη φτώχεια, την πείνα, την παιδεία, ε, την ισότητα των δύο φύλων, ε, με πολλές δηλαδή επιμέρους συνιστώσεις των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Ποιες είναι οι σχέσεις λοιπόν. Το φύλλο είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική υγεία και άρα και για τα νοσήματα. Υπάρχουν στενότατες σχέσεις με τις ε, ψυχικές ε, διαταράξεις, ε, διότι υπάρχουν κίνδυνοι που εντοπίζονται σε συγκεκριμένα φύλλα. Αν δείτε αυτό το γράφημα, παραδείγματο χάρη, βλέπουμε τη, τη, τη μελέτη. Ε, εντάξει, δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά με ε, το απαλό μπλε βλέπουμε ε, τις ε, γυναίκες που νοσούν και για την ψυχική υγεία και για, τις, για τη χρήση ουσιών πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες και επίσης είναι διπλάσιο το ποσοστό των γυναικών για την κατάθλιψη και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες διάγνωσης. Υπάρχει δηλαδή ανισότητα ακόμη και ως προς τη διάγνωση της κατάθλιψης για την εσύ και για τον τοκετό. Ε, ε υπάρχουν ναι, παραγοντές, ε, συναισθηματές, ε, παραδείγματος χαρή, άγχος, κατάθλιψη, η συνθνησιμότητα, συνθνησιμότητα για τους άντρες σχετίζεται με άλλους παράγοντες. 15% των θανάτων των μητέρων αντιστοιχούν σε αυτοκτονίες και ε, επίσης, το PTSD, ε, μετατραυματικό ε, τραύμα. Μία στις πέντε γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους είτε βιάζονται είτε απειλούνται με βιασμό. 16-50% των γυναικών γνωρίζουν κάποιο, κάποια μορφή βίας, ε, δηλαδή μία στις δύο γυναίκες, ε, αν το μεταφράσουμε σε νούμερα και βλέπουμε ότι 80% των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων ε, που πλήττονται από εσωτερικό εκτοπισμό, συγκρούσεις και ζουν σε εμπόλεμες ζώνες είναι γυναίκες. Είναι υψηλότερο ο κίνδυνο για ανάπτυξη αυτού του PTSD τη μετατραυματική ε, αγχώδου διαταραχή. Ε, ε, επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Υπάρχει διακριτική μεταχείριση για την έρευνα και χάσμα ω προ τα τεκμήρια που έχουμε. Ο καθηγητή Λουί Χαρόντε στο King's College στο Λονδίνο έχει κάνει μία μελέτη για ε, όπου καταδεικνύεται αυτή η διακριτική μεταχείριση για την έρευνα και η έρευνα που γίνεται αγνοεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τι ιδιαίτερότητε που σχετίζονται με το φύλλο, όπως έλεγε και Ρόμπιν, γενικότερα για τι ε, τις ασθένειε ασθένειες για τα θέματα υγείας. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη κατάλληλη περίθαλψη και δεν υπάρχουν ε, θεραπείες και αγωγέ κατάλληλα προσαρμοσμένε στις ανάγκες που, που νοσούν. Λοιπόν, ε, ε, πρέπει να είναι η ψυχική υγεία ε, προτεραιότητα για την πολιτική, έτσι δεν είναι. Εγώ καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Αν δούμε τι ε, ε έσκατε εξελίξει για την αναψυχική πολιτική, του βιώσιμου αναψυχιακού στόχου, παραδείγματο χάρη του ΙΕ το 2015, ε, δεν συμπεριληφθήκε η ψυχική υγεία σε αυτού του στόχου παρότι υπήρχε η σχετική εμπειρία με τις γυναίκες και για την εκπόνηση των νέων βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και όσο πλησίαζε το 2014 ε, ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι είχαμε κάνει πάρα πολλή δουλειά για να συμπεριληφθεί η ψυχική υγεία στους στόχους προέκυψε με σαφήνεια ότι μάλλον θα αποκλειστεί η ψυχική υγεία και πάλι από τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ε, ένας ε, Γάλλος ε, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ερευνητής και ψυχίατρος στο King's College, ο καθηγητής Λόνικροφτ ε, ε, αναφέρθηκε σε αυτό, είπε ότι είναι απαραίτητο και με τον καθηγητή Παντέλ στο BNC, δηλαδή στην πιο έγκυρη, στο πιο έγκυρο ιατρικό περιοδικό, απίφθηναν δημόσια έκκληση να συμπεριληφθεί η ψυχική υγεία στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ο Νίκορ Thorne Croft ε, χρηματοδοτεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση της ε, των πρωτοβουλειών για την ψυχική υγεία και τη συμπερίληψή του σε, ε, στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Έχουμε 25 διεθνεί εμπειρογνώμονες. Σε πάνω από 70 οργανώσεις μας υποστηρίζουν, ενισχύουν έτσι την παρουσία μας στο ΝΟΗΕ, ούτω ώστε να συμπεριληφθεί η ψυχική υγεία στους αναπτυξιακούς στόχους και επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Θα δείτε ένα βίντεο τώρα ε, ε, που έχει φτιάξει ο φωτογράφος Ρόμπιν Χάμοντ. <clears throat> Um, το 2014 έως το 2015 κάναμε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες ε, στον ΟΗΕ για να υποστηρίξουμε τη τη θέση μας. Ο Μίτσιν Νοχάμεν, το ειδικό σύμβολο του ΙΕ για τους στόχους, αναβιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους ε, παρά τον Μπάνκιν Μουν, ε, εξασφάλισε επίσης την υποστήριξή του και ο πρώην γραμματέας ε, του ΙΕ, Κόφι Ανάνε, είπε στο Λονδίνο ότι στα τέλη του 2014, ενώ εξετάζουμε το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο και την εκπόνηση των νέων στόχων, θα πρέπει την ψυχική γέκλωση, ιδιαίτερα στην κατάθλιψη, να τη συμπεριλάβουμε στο θεματολόγιο του 2015 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λοιπόν, ε, το 2015 πλησίαζε ο Σεπτέμβρη και δεν ξέραμε τι θα γινόταν. Από ό,τι φαινόταν θα αγνοούσαν και πάλι την ψυχική υγεία αλλά τελικά όμως προς έκπληξη όλων ε, συμπεριλήφθηκε ε, στο προήμιο επίσης της δήλωσης για του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου τονίζεται ότι συνιστά και προτεραιότητα για την εκπόνηση πολιτική ε, ε, στον στόχο 3 αναφέρεται τρεις φορές ε, για την πρόληψη και θεραπεία των διαταραχών. επίσης, στα πλαίσια της καθολικής κάλυψης για τις υπηρεσίες υγείας και για την κατάχρηση ουσιών. οι δείκτε τώρα. προτείναμε στα, σε συνδυασμό με τον ΠΟΕ και το δικτύου των ε, οργανώσεων για τους ε, αναπτυξιακούς στόχους να αναπτυχθούν δείκτες ε, για τις βασικές διαταραχές. Αυτό δεν απαιτεί κάποια περαιτέρω προσπάθεια από πλευράς των κρατών, διότι το σχέδιο δράσης του ΠΟΕ καλύπτει ήδη αυτή την πτυχή. Οι τωρινοί ε, δείκτες ε, των ε, στόχων που συμφωνήθηκαν το Μάρτιο του 2016, 230 είναι περίπου και είναι προκατακτικό βέβαια αυτό πόρισμα αυτό που σας λέω, αλλά αυτοί ε, ε, είναι οι δείκτες. Ε, παραδείγματος χάρη θνησιμότητα λόγω αυτοκτονίας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται οι σοβαρές διαταραχές. Οπότε συνεχίζουμε να πιέζουμε, να προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στον ΟΗΕ, ώστε οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές να συμπεριληφθούν αυτές καθεαυτές στους δείκτες και στους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ. Ε, ο Άιφρεντ, ένα από τα μέλη της ε, καθοδηγητικής ομάδας μας, έφτιαξε ένα νέο βίντεο και θα σας το δείξω τώρα για τον ε, αγώνα που κάνουμε στα ΜΕΓΕ. Λοιπόν, για να περάσω στα βασικά μου μηνύματα που θέλω να θυμάστε από σήμερα, η, τα ψυχικά νοσήματα ε, ε, ε, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρόκειται για ένα εγκάρσιο ζήτημα που σχετίζεται με το φύλλο, τις ιδιαιτερότητες του φύλλου. Ε, και τις πολιτικές που επονούμε Και θα πρέπει να τονωθούν οι προσπάθειες ε, στα πλαίσια των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, διότι χωρίς ψυχική υγεία και ισότητα των ευκαιριών δεν μπορούν να υπάρξουν ε, αν δεν επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Muchísimas Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βοτρούμπα. Νομίζω πως δεν έχουμε αρκετά λόγια για να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που προσπαθούν να δώσουν περισσότερη δημοσιότητα στα θέματα της ε, ψυχικής υγείας. Διότι η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχουν πολλές ε, διαβαθμίσεις. Είναι ακριβώς όπως είναι ο ήχος στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Υπάρχει ένα φάσμα. Όταν ξεπεράσεις κάποιο όριο, τότε αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους μας που έχουν ζητήσει έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τη χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, που δεν είναι και πολλοί. Η κυρία Μπιόρκ έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο ε, εισηγήτριες μας ε, και τα, μέλη του πάνελ. Όπως ξέρετε, εμείς ε, ασχολούμαστε με, πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα και με το θέμα της υγείας των γυναικών φυσικά υπάρχει και ο ε, των γεννητικών οργάνων και αυτό είναι θέμα υγείας, δηλαδή πέρα από τη ζωή είναι και ποιότητα ζωής. Ε, αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε και θα πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θα ήθελα να ακούσω αν έχετε περαιτέρω στοιχεία εσείς σε πολλά τμήματα της Ευρώπης ε, υπάρχει άνηση πρόσβαση στην ε, περίθαλψη, όχι ανάλογα με τις ανάγκες, ε, αλλά σε ε, διάφορα ε, κράτη, κυρίως λόγω της πολιτικής λιτότητας, ε, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και μην ξεχνάμε ότι πλήττει αυτό για και χώρες όπως η δική μου, τη Σουηδία, με την ιδιωτικοποίηση του τομέα της υγείας, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν ως ανώτατο στόχο το την προστασία της υγείας αλλά την αποκόμιση των ε, μέγιστων κερδών. Επίσης, ε, θα ήθελα να μιλήσω για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. 50.000 ε, γυναίκες και εκατομμύρια πεθαίνουν και εκατομμύρια παθαίνουν κάποιες μολύνσεις λόγω αμβλό, εκτρώσεων που γίνονται ε, ε, από ακατάλληλους ε, γιατρούς και φυσικά αυτό συνδέεται άμεσα με την υγεία την ζωή, το επίπεδο και την ποιότητα της ζωής και σχετίζεται φυσικά με το φύλλο. Ε, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ε, ε, τις ίσες ευκαιρίες ε, στην περίθαλψη. Όλες ε, οι γυναίκες δικαιούνται πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν γυναίκες Ρώμα και όχι μόνο οι Ρωμά αλλά και άλλες εθνικές μειονότητες, άλλες εθνότητες, μετανάστριες, φτωχές γυναίκες, οποιοδήποτε ανήκει σε μειοψηφία. Τελικά πλήττεται από αυτή την περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας σχετικές εμπειρίες, αν έχετε. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο. Ορίστε, στην κυρία Σταράς, δεν θέλετε. Και εκεί δύο θα τον πάρετε το λόγο. Όπως και η κυρία Μπιόρκ, είσαστε η κυρία Σταράς εισηγήτρια σε αυτή την ε, έκθεση που αναφέραμε προηγουμένως και ασχολούμαστε λοιπόν με τις ε, για την κλινική έρευνα και για την ψυχική υγεία. Οπότε ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Έσταρας και μετά η Σαμπρόζα. Εντάξει, Έσταρας. Παρακαλώ σύντομη και περιεκτική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπεσέρα για εισηγήτρια της συγκεκριμένης πρότασης, σημαντικότατης πρότασης για τον τομέα της υγείας και τις γυναίκες. Όταν μιλάμε για τις γυναίκες και την υγεία δημιουργούνται και έρχονται στο νου διάφορες καταστάσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στον τομέα της υγείας ή ομοιότητες ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Υπάρχουν και κοινά προβλήματα υγείας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, υπάρχουν όμως και τεράστιες διαφορές που θα πρέπει να μας κάνουν να σταθούμε ειδικότερα στα προβλήματα. Στον τομέα σαν παράδειγμα της ψυχικής υγείας το 11% του πληθυσμού παρουσιάζει καταθλιπτικά φαινόμενα και αυτό φύγει και τους άνδρες και τις γυναίκες. Από την άλλη, στον τομέα της απασχόλησης, η κατάσταση της υγείας, ε, δημιουργούνται καταστάσεις αρνητικές για τις γυναίκες διότι αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες, εργάζονται ε, μικρότερο χρόνο και παίζουν ένα μικρότερο ρόλο, δεν είναι σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων. Υπάρχει η αίσθηση σε σχέση με τους άνδρες για μη αμοιβόμενη εργασία λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν αυξάνονται και τα προβλήματα υγείας. Πάρα πολύ συχνά και η οικιακή απασχόληση δεν αναγνωρίζεται η οικιακή απασχόληση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται λοιπόν αντικείμενο αναγνώρισης και αυτό επηρεάζει άμεσα την υγεία. Αυτό επηρεάζει επίσης και το προσδόκιμο ζωής. Ζούνε περισσότερο οι γυναίκες, αλλά όχι όμως καλύτερα υποχρεωτικά. refiriéndose como buena o muy buena, 54% de ellas, cambio, Νομίζω ότι τα ποσοστά των γυναικών λοιπόν που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε προκεχωρημένη ηλικία είναι ιδιαίτερα υψηλά. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα μελετήσουμε για να δούμε ακριβώς τι στρατηγικές στον τομέα της υγείας θα δώσουν απαντήσεις. Να υπάρξει επίσης μια σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις τώρα αναπηρίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν λαμβάνονται ε, μέτρα στον τομέα της υγείας ε, να γίνεται αυτό με τη συνεργασία της ασθενούς και χωρίς την ε, σύμφωνη γνώμη του προσώπου που υποφέρει από αναπηρία να μην υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες να θέτουν σε αμφισβήτηση και την ικανότητα την οποία έχει σε νομικό επίπεδο να λαμβάνει αποφάσεις. Αντιμετωπίζουν λοιπόν οι ανάπηρες γυναίκες ε, ειδικά προβλήματα και γι' αυτό ακριβώ και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και για την Ισότητα των Ανδρών και Γυναικών ε, δεν αντιμετωπίζουν ειδικά ε, την κατάσταση την γυναικεία ή τουλάχιστον όχι με ικανοποιητικό τρόπο. las características especiales y también programas de prevención. Ευχαριστώ λοιπόν την Μπεατρίς για μια απαραίτητη έκθεση στην οποία ελπίζω να εργαστούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Εστάρας. Θα δώσω τώρα στην επόμενη ομιλήτρια το λόγο. Yes, thank you very... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, συνάδελφοι φεμινίστριες, για τις ε, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σας και τις πολύ σημαντικές ομιλίες σας. Έχουμε μια τεράστια γνώση των διαφορών και των ε, ανισοτήτων παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο φύλλα. αλλά αυτές όμως οι γνώσεις δεν μεταφράζονται σε πράξεις, δεν μεταφράζονται σε κατευθυντήριες γραμμές. Και δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τη βιομηχανία πως πρέπει να συνεργαστούμε, ούτε έχουμε καταφέρει να πείσουμε τη ιατρική για αυτές ε, τις ε, αλήθειες, για αυτή την πραγματικότητα. Πιστεύω πως χρειάζεται μια πιο συντονισμένη συστηματική προσέγγιση στην ιατρική που να συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση, την εκπαίδευση για τις ε, διαφορές και τις συνδιαιτερότητες των δύο φύλων. Χρειάζεται επίσης να κατανοήσουμε την ε, βιολογική διαφορά αυτών των ασθενειών. Διότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε εάν ένα πλάσμα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Χρειάζεται να γνωρίζουμε και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ορμονικά ε, επίπεδα, φαρμακολογία, ο, το διαφορετικό μεταβολισμό μιας γυναίκας από αυτόν ενός άντρα. Και έπειτα, σε τρίτο επίπεδο, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες ασθενείς ότι πρέπει να ρωτήσουν το γιατρό τους για το τι φάρμακα ε, μπορούν να πάρουν, πρέπει να πάρουν και οι γιατροί αντίστοιχα πρέπει να γνωρίζουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ε, δεν έχει το θέμα αυτό να κάνει μόνο με οικονομικές διαφορές, με πλούσιους και φτωχούς, ούτε μόνο με γυναίκες και άντρες. Για καταφέρουμε όμως να επιτύχουμε όλα αυτά, πιστεύω πως χρειάζεται να δημιουργηθεί ε, κάτι σαν ένα πειθαρχικό συμβούλιο για ε, την ε, ιατρική, για τους γιατρούς, το οποίο θα ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Θα υιοθετήσει μία ολιστική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει και την έρευνα, και την ε, βιολογία αλλά και θα τη συνδυάσει με την ε, συμπεριφορά βιολογική και μη των ε, ανθρώπων, των γυναικών. Χρειάζεται λοιπόν όσοι ασκούν ιατρικά επαγγέλματα να έχουν επαρκή κατάρτιση. Χρειάζεται όμως και επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση για τα παιδιά από νωρίς, από το σχολείο θα μπορούσε ίσως να είναι και ένας κλάδος πανεπιστημιακών σπουδών. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα από τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να αρχίσει η ευαισθητοποίηση από τη βάση και όχι από την κορυφή, έτσι όπως προσπαθούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από, τη, από το επίπεδο των ε, πολιτικών. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι ώστε η ισότητα άντρων και γυναικών να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Την τόσο επεξηγηματική θα έλεγα. Επεξηγήσατε το προφανές βέβαια. Πραγματικά ότι θα είναι, είναι περίεργο ότι αναγκαζόμαστε να εξηγούμε το προφανές πλέον. Να πούμε ότι πράγματι θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις ομοιότητες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε λίγα λεπτά στο τέλος, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συγκεκριές μας να απαντήσουν δεν θα μπορέσω να δεχθώ περισσότερες ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μορβάη, η οποία έχει ζητήσει ήδη το λόγο. Να τη ζητήσω παρακαλώ να είναι αρκετά σύντομη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ μια ομάδα επισκεπτών, παιδιά, αθλητές του handball από την Ουγγαρία. Πιστεύω πως πρέπει να μας θυμίζουν πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός ε, σε αυτά που συζητάμε σήμερα. Όχι μόνο δηλαδή σημαντικός για την διατήρηση της ψυχικής υγείας, αλλά και για την αποκατάσταση μιας κλονισμένης ψυχικής υγείας. Όπω είπε η πρώτη ομιλήτρια, αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι οι καρδιακιακέ παθήσει είναι το κύριο αίτιο θανάτου ε, για τις γυναίκες. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που ε, αφορά πολλά κρατημέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου. Οι γυναίκες είναι οι υπεύθυνε ακόμα και τώρα για ε, των οικοκυριών. Κάνουν δουλειέ του σπιτιού, φροντίζουν ηλικιωμένου, φροντίζουν μέλη της οικογένεια και πρέπει ταυτόχρονα να είναι σωστέ επαγγελματίε. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε που αντιμετωπίζει μία γυναίκα έτσι ώστε ε, πολλές από αυτές παραμελούν την υγεία τους, παραμελούν ε, την σωματική υγεία τους, δεν αθλούνται. Τι θα, μπορούμε, λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε για να αλλάξει αυτό, για να βελτιωθεί η θέση των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με την κυρία Μπότροβα και αμέσως μετά με την κυρία Νόρτον. Παρακαλώ δύο λεπτά η καθεμία από σας. Ίσως να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις παρατηρήσεις οι οποίες σας αφορούν ή να βγάλετε κάποια ίσως μικρά συμπεράσματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο κινούμεθα στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι αποκαλυπτικό ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε όπως θα έπρεπε, δεν τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, από δύο λεπτά η κάθε μία από εσά για να απαντήσετε και να κλείσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Μπότοβα, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία πολλοί αναφέρονται σε αυτά τα οποία είπα στην παρουσίασή μου. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται από την κυβέρνηση στον τομέα της πρόνοιας θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα λοιπόν φροντίδας και στον τομέα της ψυχικής υγείας και υγιεινής. Τίθενται λοιπόν προβλήματα και σε επίπεδο σχεδιασμού των πολιτικών αυτών και της παρέμβασης της πολιτικής γενικότερα, αλλά όπως είπατε ήδη, κάποια από τα θέματα αυτά ήσαν γνωστά, αλλά παρότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλά δεδομένα για τις ψυχικές ασθένειες και ειδικότερα για τις ψυχικές ασθένειες των γυναικών, εν πολύ αγνοούνται παρά το ότι ε, η αυτοκτονία είναι ε, σε καθοριστική θέση, ιδιαίτερα για τις μικρές ηλικίε. Απαιτούνται λοιπόν μεγαλύτερες και περισσότερες έρευνες, η ανάγκη είναι σαφής, πρέπει να ψάξουμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερες μελέτες και για να την αντιμετώπιση των ανισοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν τους άνδρες από τις γυναίκες, σαν παράδειγμα οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες ή είναι σε ηλικία τεκνοποιίας δεν ε, μπορούν να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές. Οπότε εδώ έχουμε ένα θέμα αν χρειαστεί τέτοιου είδους ηλικίες να τις ε, βοηθήσουμε σε ιατρικό επίπεδο. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα όπως ε, η φροντίδα ή μάλλον η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ε, και στον τομέα της ψυχικής υγείας ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια της οικιακής βοήθειας η οποία δίδεται σε ορισμένες κατηγορίες γυναικών Θα πρέπει λοιπόν η ψυχική ιδία να εγγραφεί στον κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συνδρομή αν δεν υπάρχουν προσπάθειες και στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπως είπε και η συνάδελφος από την Ουγγαρία, το θέμα τίθεται και στον τομέα των ψυχικών παθήσεων. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αντιμετωπίζουν την δυνατότητα ανάπτυξης και παθολογικών σωματικών αριθμιών πολύ υψηλότερη από ότι οι υγιείς ψυχικά συμπολίτες τους. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ κύριε Μποτρόβα. Χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Έλεγα λοιπόν στην Ισπανία ε, λέγεται ότι κανείς δεν έχει περισσότερο δίκαιο από ότι ο Άγιος αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι τα θέματα αυτά όλοι τα γνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά όλοι τα αναγνωρίζουμε είναι προφανέστατα είναι προφανές ότι η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της παροχήν υπηρεσιών. Δεν υπάρχει τίποτα το ανθρώπινο το οποίο να μην είναι σωματικό. Δεν υπάρχει τίποτα το ανθρώπινο το οποίο να μην είναι ψυχικό. Θα λόγω λοιπόν το λόγο στην κυρία Νόρτον. Δεν θέλω να κλέψω το χρόνο της. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που κάνατε και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την συνάδελφο που αναφέρθηκε στην ιατρική και τη διαφορά στα δύο φύλλα. Θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσω το πόσο σημαντική είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών γίνεται κάπως ε, κάθετα. Θα δώσουμε φάρμακα γι' αυτό, γι' αυτό και γι' εκείνο. Όχι, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Είναι πολύ σημαντικό σίγουρα να συνεργαστούμε με ε, της ε, των γυναικών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Είναι όμως επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε για την ψυχική ε, υγεία. Ξέρω για παράδειγμα ότι στην Κίνα πολλοί συνάδελφοι μου λένε ότι οι γιατροί συνιστούν στις εγγύους να σταματήσουν οποιαδήποτε ε, αθλητική δραστηριότητα. Να μην ε, κινούνται πολύ, να μην αθλούνται. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να δούμε πώς μπορούμε να εθετήσουμε μια ολιστική ε, προσέγγιση. Έπειτα, βλέπουμε πώς πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις ε, βασικές διαφορές και το πώς αυτές μεταφράζονται σε, στην υγεία. Τέλος, περικοπές στον ε, χώρο της υγείας. Σίγουρα χρειάζεται να μειωθεί το κόστος, όμως αυτό ε, μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται να είμαστε λοιπόν πιο δημιουργικοί, πιο καινοτόμοι για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με διάφορους ε, τρόπους, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουμε ε, διάφορους επαγγελματίες υγείας που δεν είναι ε, απαραίτητα οι γιατροί, να δούμε πώς μπορούμε δηλαδή να διατηρήσουμε την υγεία εκτός το, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έπειτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και το ιατρικό ερευνητικό συμβούλιο, το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζει τις διαφορετικές δυνατότητες που έχουμε ε, ως προς τη χρηματοδότηση. Μία από αυτές τις δυνατότητες που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι χρηματοδότηση για ε, θέματα ε, που αφορούν τα δύο φύλλα. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν μπορώ να αλλάξω αυτά που ήδη έχουν γίνει. Μπορώ όμως να κάνω τη διαφορά για αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία των υπεύθυνων ε, για την ε, χάραξη πολιτικής. Το θέμα του φίλου είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές ακόμα και άτομα όπως εγώ που ασχολούμαστε όλοι μας στη ζωή με αυτό ξεχνάμε να συνεκτιμήσουμε τη διάσταση του φίλου σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση και ξέρω πως ακούγομαι ε, βαρετή, ίσως πως επαναλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά θέλει προσοχή. Σας ευχαριστώ κυρία Νόρτον. Νομίζω ότι όλοι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τέτοιου είδους συζητήσεις ε, όχι μόνο είναι θετικές αλλά μπορεί να είναι η πραγματική αιτία και ο λόγος των αλλαγών. Πολλές φορές οι αλλαγές ε, εξαρτώνται από μια απλή πολιτική απόφαση. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή το αναγνωρίσουμε τότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να προκαλέσουμε τις ίδιες τις αλλαγές. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στην κυρία Νταμόνσε έτσι ώστε να βγάλει και αυτή τα δικά της συμπεράσματα πριν περάσουμε στο επόμενο πάνελ. Just in closing. Ναι, να κάνω κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Νικόλ, ευχαριστώ καθηγητή Νόρτον. Νομίζω ότι μετά από αυτό το πάνελ Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το, είναι το φύλλο για τις μη μεταδεδόμενες ασθένειες και την ε, ψυχική υγεία. Ε, και δεν είναι αυτό τόσο γνωστό, δεν ακούγεται πολύ. Ε, Νόρτον, ε, πολύ σωστά μας είπατε ότι εστιάζουμε στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και όλα τα συναφή ζητήματα. οπότε καλό είναι που το ακούσαμε σήμερα στο πάνελ μας. Κάποιες από τις ιδέες που ακούσαμε. Αυτές οι μη μεταδεδόμενες ασθένειες και η ψυχική υγεία δεν συνδέονται μόνο με το στυλ διαβίωσης των ε, πλουσίων και διασύμων. Το μεγαλύτερο βάρος το φέρνουν οι φτωχές χώρες ε, πέρα από τα μεταδιδόμενα νοσήματα φέρνουν το μεγαλύτερο βάρος και υπάρχουν, είναι ο μεγαλύτερος επιπολασμός σε αυτές τις χώρες για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και για τις διαταραχές ψυχικής υγείας. Σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι θέματα των χωρών ε, υψηλού εισοδήματος. Όχι, αυτό δεν ισχύει ε, και αποδεικνύεται από τα στοιχεία που είδαμε και άρα θα πρέπει για την ζωή και την ποιότητα της ζωής να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, μας μιλήσατε για τις πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα των ε, γυναικών. Θα πρέπει να γίνεται μαστογραφία ε, ή τεστ παπ ή τσεκάπ μία φορά το χρόνο για τον καρκίνο, για τις καρδιακές παθήσεις. Οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου, πώς λειτουργεί ο είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, γίνονται δράσεις ευαισθητοποίησης των γυναικών. Για την ενσωμάτωση, αναφέρθηκε αυτό στις περισσότερες ομιλίες. Ολιστική προσέγγιση χρειαζόμαστε, όχι μόνο βιολογική, πρόπτικη, προοπτική, ε, το, των ζητημάτων. Όχι, υπάρχει τα, τα οικονομικά ζητήματα, τα κοινωνικά ζητήματα, όλα αυτά σφαιρικά θα πρέπει να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Η προσέγγιση επίσης για τα δευτερογενή στατιστικά δεδομένα μετά την έρευνα. Θα τα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα από αυτό το φακό ε, των, ε, της ισότητας των δύο φύλων. Στο προηγού, στην προηγούμενη σύνοδο αυτό ήταν από τα βασικότερα συμπεράσματα. Δηλαδή η Παγκόσμια Οργάνωση Χρηματοδότη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια τέτοια συνολική προσέγγιση και γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα δευτερογενή φιλτραρισμένα μέσω του φύλου στατιστικά δεδομένα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ζήτημα των νέων προσεγγίσεων για την έρευνα δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Σήμερα το πρωί νομίζω ότι αυτό μας αποσχόλησε κυρίως, να μην απολαμβάνουμε τα ίδια, να υιοθετήσουμε κάποιες πιο ρηξικέλευτες προσεγγίσεις όπως αυτές που προτάθηκαν σήμερα το πρωί για την έρευνα. Έτσι μπορούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τις συζητήσεις μας για την επόμενη μια μισή μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συζητήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Νόρτον, ευχαριστώ την κυρία Μποτρούβα. Μια σκέψη θα ήθελα και εγώ να κάνω, λέει η Πρόεδρος. Μια και εδώ είμαστε εκπρόσωποι της Λαϊκής Βούλησης και εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων είναι σαφές ότι δεν έχει, λένε ορισμένοι ότι δεν έχει αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχει αρμοδιότητες στον τομέα της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει αρκετές εκθέσεις και για τον ρόλο των γυναικών και τη θέση των γυναικών. Το θέμα είναι ότι τα έγγραφα αυτά δεν έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα πολιτικά προγράμματα για βελτίωση των, της θέσης των γυναικών στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Έχουμε λοιπόν αρμοδιότητες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μελέτες κατάλληλες, πολιτικά μέτρα, παρεμβάσεις, αποφάσεις εναντίον των λαθών και των διακρίσεων δεν έχουμε. Πρέπει να τις αποκτήσουμε. Πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν η προοπτική της ισότητας των φύλων να χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν παράδειγμα στον τομέα της υγείας δεν χρηματοδοτείται η έρευνα σε ό,τι έχει σχέση με την υγεία και την προβληματική των φύλων. Αυτά είναι θέματα τα οποία αποσχαλούν και την έκθεση με την οποία σε αυτή την εποχή στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική των Γυναικών. Νομίζω ότι με προσπάθειες, με περαιτέρω έρευνα θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις με βάση το φύλλο. Είναι άδικο, είναι κάτι το οποίο συνιστά διακριτική μεταχείριση, είναι αναποτελεσματικό και είναι πάρα πολύ κακό για την πρόοδο, για την ανάπτυξη, για την οικονομία. Πρέπει να αλλάξει γιατί δεν μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε τον βασικό μας στόχο που είναι η ισοτιμία ανδρών και γυναικών. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους που μας συνέδωσαν μέχρι τώρα. Λυπάμαι που δεν έδωσα το λόγο σε όλους όσους το ζήτησαν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν προχωρήσουμε να ευχαριστήσω την κυρία Μπότρουβα και την κυρία Νόρτον και θα διακόψουμε για ένα-δύο λεπτά.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 Good morning. Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ να καθίσετε, λέει η κυρία Βόζεμπερκ, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να με ακούσετε. Can't you listen? Does it function? You can, you can listen to me. Υπάρχει προφανώς ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λύθηκε όμως. Σας ευχαριστώ, λέει ξανά η κυρία Βόζεμπερκ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Η σημερινή μας συνάντηση. Το αντικείμενο της ημερίδας μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και λίγων μόνο, με λίγα λόγια, να σας πω ότι είχα την τιμή πέρσι να είμαι εισηγήτρια σε μια έκθεση για την γυάλινη οροφή, το glass ceiling όπως λέγεται, και το οποίο σημαίνει ακριβώς εκείνα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καριέρας που απευθύνονται σε τομείς στο ανώτατο επίπεδο στην έρευνα στο πανεπιστήμιο στην τεχνολογία και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι γυναίκες αυτές, αλλά και οι δρόμοι που ακολουθούν αντιμετωπίζουν πόδια από κάποια στερεότυπα που θέλουν να προτιμώνται οι άντρες ακριβώς σε αυτές τις, θέσεις, ε, τις ανώτατες θέσεις καριέρας. Η σημασία του να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη, σε μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική, έγκυται στην γνώση ότι οι γυναίκες που υπηρετούν τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς που προαναφέρθηκα, δηλαδή στην έρευνα, στην τεχνολογία, στο πανεπιστήμιο, συμβάλλουν καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, συμβάλλουν καθοριστικά στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι επαρκής για την αναγνώριση των γυναικών και των δικαιωμάτων των γυναικών να έχουν εκείνα τα κίνητρα ώστε να επιδιώκουν τους ύψιστους στόχους, έχουμε δει ότι στην πράξη αυτό τελικά δεν τηρείται. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη. Και ο δρόμος αυτός περιλαμβάνει και την ανάγκη εξέλιξης και της νομοθεσίας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών ξεχωριστά. Ερχόμενοι στην αίθουσα θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο έχει μια ε, δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μας στην ε, γυάλινη οροφή, αλλά δείχνει παγιωμένες νοοτροπίες εναντίον των οποίων εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα και στις προσπάθειές μας μέσα από την Επιτροπή Γυναικών παλεύουμε. Θα δείτε αναρτημένους τους διαδρόμους τους παρελθόντες προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους τρέχοντες των τρεχόντων ετών μέχρι σήμερα. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι 28 άντρες μεταξύ των οποίων μόνο δύο γυναίκες. Αυτό και μόνο αντιλαμβανόμαστε ότι δείχνει μια ανισότητα, διότι κανένας δεν πιστεύει ότι ανάμεσα ε, μεταξύ αυτών των 28 θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχα 28 γυναίκες με τα ίδια προσόντα, με τις ίδιες ικανότητες, με παραγωγική σκέψη και με σκληρή δουλειά. Έτσι λοιπόν, ε, κάνοντας αυτή την ε, έναρξη, εναρκτήρια εισαγωγή στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι οι γυναίκες καριέρας θα πρέπει όχι μόνο να μην βρίσκουν εμπόδια, αλλά αντίθετα με παγιωμένες, ολοκληρωμένες νομοθεσίες στα κράτη-μέλη και μια ολοκληρωμένη, οριζόντια αλλά και σφαιρική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκουν κίνητρα έτσι ώστε να ενθαρρύνονται, να επιτυγχάνουν το στόχο τους, διότι έχουν αποδείξει ότι σήμερα Ευτυχώς δεν υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα, γυναικοί και ανδρικοί στόχοι. Υπάρχουν στόχοι τους οποίους κάθε άνθρωπος μπορεί ανεξαρτήτως φύλου να τους επιδιώκει, να οργανώνεται και με μεθοδική δουλειά να τους επιτυγχάνει. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Elizabeth Πόλιτζερ. She's co-founder and director of Portia στον τομέα των STEM, στον τομέα δηλαδή μαθηματικών τεχνολογίας και μηχανικής, για τα STEM μιλάμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο ισότιμη είναι η πρόσβαση των γυναικών στα STEM. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και έχω την αίσθηση πως βρίσκομαι εδώ ε, μπροστά σε μια κοινότητα η οποία ολοένα και μεγαλώνει από το 2011 που έγινε η πρώτη μας ε, σύνοδος. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών που έδωσε τη δυνατότητα στην ε, σύνοδό μας να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2012 συζητούσαμε τον ορίζοντα 2020 εδώ και αυτή η συζήτηση επηρέασε πάρα πολύ σημαντικά τις εξελίξεις και το πώς η ισότητα των φύλων συμπεριλήφθη στο πρόγραμμα αυτό. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε πώς ε, η συνεργασία ανάμεσα στην πολιτική και στους ε, επιστήμονες και στους πανεπιστημιακούς μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις για τις ε, γυναίκες. Στόχος ε, λοιπόν σήμερα είναι να δούμε τι γίνεται στις άλλες περιοχές του κόσμου όπου η σύνοδος αυτή που κάνουμε σήμερα χρησιμοποιείται έτσι ώστε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα για τις ανάγκες των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πόλιτσαρ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μιγιώκο Βατανάμπε. Ελπίζω να προφέρω καλά το όνομά σας. Αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια για την ε, Υπηρεσία Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Θα μας μιλήσει για την πολυμορφία και την ε, χωρίς αποκλεισμούς Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σα μιλήσω για την επόμενη σύνοδο στην Ιαπωνία και το τι κάνουμε εμεί. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με πολλού έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα στην Ανατολική Ασία. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βλέπετε εδώ την ιστορία της διασκεψής μας. Η επόμενη διάσκεψη θα γίνει στις 25 και 26 Μαΐου του 2017 ε, σε μία αίθουσα που βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό του Τόκιο και βολεύει λοιπόν στις μετακινήσεις. Επόμενη διαφάνεια, η δομή των επιτροπών μας. Εδώ βλέπετε τη δομή του δικού μου οργανισμού και του Συμβουλίου δηλαδή Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. συνεργαζόμαστε με την ε, Ακαδημία της Ιαπωνίας για πολλά θέματα. Έχουμε τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων όπου, όπως σας είπα, αναφερόμαστε σε διάφορα πολύ σημαντικά θέματα για τις ε, γυναίκες. Επίσης, ε, έχουμε διάφορους ε, συμβούλους οι οποίοι μας ε, παρέχουν μεγάλη βοήθεια στο έργο μας. Έπειτα, το Συμβούλιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς και με, την, με τον οργανισμό Πόσια, αλλά και με πολλά υπουργεία της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και επαγγελματικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε επίσης και με δύο πανεπιστήμια της Ιαπωνίας και ε, με έναν οργανισμό καινοτομίας της Κορέας. Επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς, περισσότερα ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και να διευρύνουμε τη βάση των ε, χορηγών μας. Αυτή τη στιγμή οι χορηγοί μας είναι αυτές οι 8 εταιρείες που βλέπετε στην ε, διαφάνεια. Τρία πανεπιστήμια, 16 πανεπιστήμια στην Ασία. Έχουμε δηλαδή 26 χορηγούς στο σύνολο. Ελπίζουμε να επεκταθούμε και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τη δομή της χορηγίας. Έχουμε τρεις μορφές χορηγίας. Και σημαντικό για εμάς είναι να αποκτήσουμε περισσότερους ε, διεθνείς εταίρους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, ζητήσω, αν ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγοί, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θέμα τώρα της έσκεψης είναι καλύτερη επιστημονική καινοτομία και συμπερίληψη των γυναικών. Σχεδιάζουμε τρεις ολομέλειες. Στην πρώτη θα συζητηθούν τα σύνορα, τα όρια του ταλέντου και το πώς μπορούμε να επεκταθούμε σε όλους τους τομείς των επιστημών. Θα συζητηθεί επίσης το θέμα της προσβασιμότητας και της ε, τεχνολογίας των ε, διεπιφανειών. Έπειτα, θα συζητηθούν επίσης διάφορες ε, προτεραιότητες που έχουν κυρίως οι ασιατικές χώρες. Θα συζητηθεί επίσης το θέμα της έλλειψης τροφίμων, της πείνας, της φτώχειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην τρίτη Ολομέλεια θα συζητηθεί το θέμα της κοινωνικής ευθύνης της ε, επιστήμης, του επιστημονικού κλάδου. Η κυρία Χιαγιάμα θα προεδρεύσει από το Επιστημονικό Επιμελητήριο της Ιαπωνίας. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια τους ε, υπόλοιπους καλεσμένους μας. τον, την Dr. Πικ που βλέπετε εδώ, που μίλησε και νωρίτερα. Θα συζητηθεί λοιπόν η κοινωνική ευθύνη της επιστήμης. Θα γίνουν επίσης και δύο σχετικά συνέδρια και να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο κατάρτισης προτάσεων για το περιεχόμενο της 10ης διάσκεψης Gender Summit 10. Στόχος μας είναι να συζητηθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να καλύψουμε μόνο τους 5 από τους 17 στόχους. Θα συζητηθούν λοιπόν θέματα τα οποία αφορούν το φύλλο, ε, τους νέους ανθρώπους, τα γόρια, τα κορίτσια, της, ε, τη μητρότητα. Αυτά τα θέματα καλύπτουν τα δύο τρίτα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Τώρα, στα αριστερά αυτής της διαφάνειας βλέπετε τους στόχους που συνδέονται με το φύλλο. Και στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας βλέπουμε τους στόχους οι οποίοι δεν ε, συνδέονται με το φύλλο, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση των στόχων αυτών με το φύλλο. Στόχος είναι αυτοί οι στόχοι να φορούν εξίσου άνδρες και γυναίκες. Όμως, πολλοί από αυτούς τους στόχους αφορούν και τη βιομηχανία. Αυτό τι μας λέει. Μας λέει ότι η βιομηχανία πρέπει να ασχοληθεί με τη διάσταση του φύλου, διότι εάν θέλουμε να έχουμε επιτυχία και να καταφέρουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να γίνει αυτή η συνεκτίμηση της διάστασης του, του φύλου σε όλους τους στόχους. Εδώ βλέπετε τον ιστότοπό μας, μπορείτε να τον επισκεφθείτε και να σας ενημερώσω για τις εγγραφές. Θα αρχίσουν στις 28 Νοεμβρίου και η καθηγήτρια κυρία Κουμινόσε θα σας μιλήσει για τις λεπτομέρειες ε, της... Ε, διάσκεψης αυτής. Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει κυρία Βοζενπέκ. Έχουμε όμως πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Ινώσε τώρα είναι αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ε, Ιαπωνίας και καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια. Ε, το, για τη σύνοδο που θα γίνει την επόμενη χρονιά θα ηγηθώ δύο ε, προ, πάνελ ε, προπαρασκευαστικών για να δούμε τις τελευταίες τάσεις σε σχέση με τα ζητήματα που σχετίζονται με τα δύο φύλλα. Βλέπετε την ημερίδα που έγινε το 2014 στο Ελσίνκι ε, να ηγηθείτε της αλλαγής, να είσαστε η αλλαγή. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ο στόχος όλων των κυβερνητικών οργάνων θα πρέπει να είναι μέχρι το 2020 40% εκπροσώπηση <laughs> των γυναικών και μιλούμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ε, τρίτο ε, σημείο, εκεί είχαμε δύο διαφορετικά πάνελ πρώτον για τις επιδόσεις των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την ισότητα των ευκαιριών στην κοινωνία. Με αυτά τα στατιστικά δεδομένα βλέπουμε πως σχετίζεται ε, το φύλλο με τις επιδόσεις των γυναικών και ξαναλέω αυτό ε, αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 ε, στο Τόκιο. οι αθλήτριες λοιπόν ήταν το αντικείμενο της έρευνας από 44 ε, χώρες ε, χρησιμοποιώντας ε, το GTI, το δίκτυ GTI. στη συνέχεια εξετάζουμε, περάστηκε στην επόμενη διαφάνεια, το, θέμα των ειδικών αναγκών πέρα από τη, τις τα ζητήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες ε, θα πρέπει να περάσουμε, να εξετάσουμε και τα πολιτισμικά ζητήματα, τα θέματα κουλτούρας ε, και νοοτροπίας, ε, θέματα ανταγωνιστικότητας για την, μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες παραδείγματος χάρη μπορούμε να αναπτύξουμε μια διαφορετική νοοτροπία, μια νέα κουλτούρα. Στη συνέχεια, εξετάζοντας το θέμα από την οπτική γωνία των αντρών. Βλέπουμε βάσει της πρόσφατης αυτής μελέτης ε, ότι για τις, ε, για τις επιστήμες ε, τελικά έχουν καλύτερες επιδόσεις τα κορίτσια και οι γυναίκες. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 στην Ευρώπη βεβαιώνεται αυτή η τάση. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα αυτών των επιδόσεων που διαπιστώνεται ανά τον κόσμο και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε τα στατιστικά δεδομένα ε, στα φύλλα. Η Μιώκο και εγώ συνεργαζόμαστε στενά για να προετοιμάσουμε την ε, δέκατη σύνοδο για, για το φύλλο ε, και σας περιμένουμε όλους στο Τόκιο. Σας ευχαριστούμε. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Λή, ε, βασική ερευνήτρια στο ε, Κέντρο Ερευνητικής Καινοτομίας ε, Τσίρκ. Παρακαλώ. να μιλήσω λίγο αναφερόμενο στα θέματα της καινοτομίας. Ο συσχετισμός της καινοτομίας συμπεριελήφθη στο τρίτο πρόγραμμα για την προώθηση της θέσης των γυναικών στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Τα θέματα της εφαρμογής της προβληματικής των φύλων στην έρευνα συστηματικά ενσωματώθηκε στην Κορέα στην προετοιμασία της συνάντησης κορυφής ε, της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Κορέα το 2015. Από εκεί που φροντίζαμε μόνο τα ποσοτικά στοιχεία, τώρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά θέματα που προκαλούν αυτές τις διαφοροποιήσεις Βασιζόμενοι λοιπόν και στα δεδομένα και στην πολιτική συμπερίληψη των γυναικών, το ερευνητικό, δημιουργήθηκε το ερευνητικό κέντρο το Δεκέμβριο. Έγινε και μία συνάντηση κορυφής για τα φύλλα το 2015 για την επίτευξη της ισότητας και την συμπερίληψη της προβληματικής των φύλων μεταξύ ε, δε άλλων θεμάτων και το θέμα της καινοτομίας. Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές για την εφαρμογή κάποιων από αυτές τις καινοτομίες. Το NRF το ερευνητικό ίδρυμα της Κορέας στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Το Ίδρυμα Έρευνας λοιπόν The next slide, please. The Gender Summit. Η συνάντηση κορυφής λοιπόν για τα φύλλα αναφέρθηκε στους στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών. Έγιναν πολλές αναφορές για την συνεργασία με τις υπηρεσίες των Μένων Εθνών, όπως το δίκτυο αηφορίας και επίσης συνεργασία υπήρξε και με τον ΩΣΑ, έτσι ώστε να κατατεθούν προς τα απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα. Το Τζίστερ έκανε έρευνες και σε επίπεδο προσπάθειας των ορισμών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του πεδίου δράσης στην Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετατραπεί η πολιτική αυτή σε συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της νομοθετικής ρύθμισης για την έρευνα και την τεχνολογία βασικός στόχος του Τζίστερ είναι να προωθήσει λοιπόν την καινοτομία και στις, τα προγράμματα διδασκαλίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και σε επίπεδο χρηματοδότησης. Το Τζίστερ μέχρι τώρα έχει ολοκληρώσει κάποιες κατά περίπτωση μελέτες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Λέγοντας σε ποιο βαθμό Research covers basic science, biomedical research, engineering, environment. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό σχετικά το επίπεδο στο οποίο έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Η επόμενη διαφάνεια. Το κέντρο συνεργάζεται με επιμέρους οργανώσεις όπως με την Κορεατική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών που έχει κεφτεί ένα πρόγραμμα καινοτομιών για την τέταρτη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις αλλά κάναμε μια καλή νομίζω αρχή. Μια άλλη μορφή συνεργασίας είναι με την ε, ε, Επιτροπή Εκπαίδευσης στον τομέα της μηχανικής. Θα συνεχίσει η Κορέα τις προσπάθειες για να βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. you Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλήγουμε τώρα στον μόνο άντρα προσκεκλημένο, τον κύριο Σέρις Βιλεμούρ, από το Ερευνητικό Συμβούλιο Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής. Έχετε το λόγο. Μπορούμε να αρχίσουμε με τη δεύτερη διαφάνεια, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ξύπ, Πρόεδρε, Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να εκφράσω τι θερμότατε ευχαριστίε μου για την πρόσκληση στην ε, διάσκεψη για το φύλλο. Θα ήθελα να σα δώσω την ε, άποψη του δικού μα Ινστιτούτου του Καναδά. Θεωρούμε πως η διάσκεψη είναι ένα πραγματικό ε, γεγονός που βοηθά να συνδέσουμε και να μάθουμε πληροφορίες, να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μας χαρά είμαστε εδώ. Η Μαρή Κιουρί είχε πει κάποτε ότι μου έμαθαν ότι η πρόοδος δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε εύκολη και αυτό πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας συνοδεύει στις αναζητήσεις μας και στις προσπάθειές μας. Δεν θα είναι λοιπόν ούτε εύκολο ούτε γρήγορο να προχωρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να καταλάβουν την επιχειρηματική πτυχή της ε, διαφορετικότητας ε, των δύο φύλων. Η πραγματικότητα είναι ότι το κυρίαρχο μοντέλο αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και αμφισβητείται επίσης και η κυρίαρχη κουλτούρα. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι είμαστε προκατηλημένοι και ότι σίγουρα μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις. Πολλές βελτιώσεις στον ερευνητικό χώρο, στην πολιτική και την κατάρτιση αυτής. Είναι όμως μια διαδικασία που γίνεται σταδιακά και μαθαίνουμε κάνοντας. Χρειάζεται επίσης προσοχή και χρειάζεται να είμαστε επικοδομητικοί. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε για την διαφορετικότητα των φίλων και για την ισότητα άτομα τα οποία θεωρούν πως δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έτσι πάμε ένα βήμα προς τα εμπρός στην ε, πλήρη υλοποίηση και ενσωμάτωση της ισότητας. Έπειτα πρέπει να συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να ενημερώνουμε βασισμένοι σε στοιχεία. Ας δούμε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα, με τα οχήματα. Είναι αυτή τη στιγμή ε, επικίνδυνα και τα τροχαία ατυχήματα είναι μία από τις ε, κυριότερες αιτίες θανάτου βρεφών και εμβρίων. Μετά, μία έρευνα που ε, διεξήχθη από το Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών του Καναδά ε, είναι πιστεύω πάρα πολύ χρήσιμη, έχει πολλά γραφικά και μπορούμε να την κατανοήσουμε. Ε, μπορούμε να δούμε μέσω της έρευνας αυτής τι συμβαίνει με την διαφορετικότητα των δύο φύλων. Αυτά λοιπόν εν συντομία και θα δώσω το λόγο πάλι σε εσά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τώρα το λόγο στον κύριο. Κυρία Μαρίς Λασόντ από το Επιστημονικό Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Καναδά. Έχετε το λόγο. Χαίρομαι που είμαι εδώ και θα σας μιλήσω για την 11η σύνοδο που θα γίνει στο Κεμπέκ. Ο Πρωθυπουργό μας, ε, ο Καναδάς, έτσι τα αναγνωρίζετε και πέρσι μας ρώτησαν γιατί είναι σημαντικό ε, να έχετε ισότιμη εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί είναι το 2015, ελπίζουμε το 2017 θα φέρει Ισότιμη εκπροσώπηση. επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε διάφορα παραδείγματα πρωτοβουλίων στρατηγικού σχεδιασμού και μεταξύ άλλων για την ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε την Gender Present Analysis Plus. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου για το καθεστώς των γυναικών. Ε, είναι, όπως είπαμε, πρωτοβουλία του Υπουργείου και το Ινάριο του 2017 για ε, το Εθνικό Ινστιτούτο για την έρευνα στη μηχανική και στις φυσικές επιστήμες ε, προσυπέγραφει επίσημα αυτή την πρωτοβουλία για την ισότητα των δύο φύλων και ασχολείται και με την εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης δέσμευσης. Το FRQND είναι ε, το Ινστιτούτο στην επαρχία του Κεμπέκ, ε, όπου είμαι πρόεδρος και σε συνεργασία με την UNESCO θέλουμε να μετάχουμε στο πρόγραμμα ε, για την προώθηση της ισότιμης εκπροσωπής των γυναικών στις θετικές επιστήμες ε, εστιάζοντας στη μηχανική στα μαθηματικά στις ε, θετικέ επιστήμες, το GenderNet, αυτό είναι για την Ευρώπη φυσικά και η διεθνή Πρωτοβουλία για την Έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτή τη πρωτοβουλία. Επόμενη διαφάνεια. Ε, Αυτά είναι από, το προηγούμενο, από την προηγούμενη σύνοδο, το Παγκόσμιο Ερευνητικό Συμβούλιο, παραδείγματο χάρη. Εφαρμόζουν κάποια σχέδια δράσης ερευνητικά, ένα εν είδη παραδείγματος, ε, ερευνητικές ευκαιρίες ε, για τις γυναίκες που δεν μπορούν να δημοσιεύσουν διότι έχουν άδεια σε ποιε είναι οι δυνατότητε έρευνα, ε, έχουν αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, διαπιστώθηκε ανάλυση ε, σε σχέση με το φύλλο, επίσης, ε, το Ερευνητικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και παραθέτω λέει ότι η παρεκβολή των αποτελεσμάτων σε ολόκληρο ε, το πληθυσμό ε, είναι παραπλανητικό και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε παγκόσμια στοιχεία και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να συμμετάσχουμε και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο και στο Gender Summit. Επόμενη διαφάνεια. Στο 10ο, στη δέκατη Σύνοδο Κορυφής έχουμε τέσσερες βασικές ομάδες ποικιλομορφία στην λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις, ε, στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και στην έρευνα. Επίση θέλουμε να επιτύχουμε διασυνδεσιμότητα κατά το στήριο 50 επέτειο και <clears throat> θέλουμε διασυνδεσιμότητα και με τον κόσμο πλουραλισμός, ε, ε, αυτόχθονες πληθυσμοί, ε, ενσωμάτωση των φύλων, ισότητα των δύο ευκαιριών. Φυσικά είναι μια πληθυσμιακή ομάδα στον Καναδά οι αυτόχθονες που δεν εκπροσωπούνται στην έρευνα και πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, για την Βόρεια Αμερική θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους οργανισμούς, ώστε να αποκτήσουμε διεθνή παρουσία. αυτή. είναι βασικά ερωτήματα, κάποια από τα βασικά ερωτήματα που ε, συζητάει η περιφερειακή διάσκεψη εν ώψη της Συνόδου 11 που θα γίνει στο Μόντρεαλ όπως σας είπα σε ένα χρόνο από τώρα ε, τα ζητήματα που πραγματευτήκαμε στην προηγούμενη σύνοδο τι θέλουμε να επιτύχουμε με αυτή τη νέα σύνοδο ε, πώς ε, να μεταφραστούν το αποτελέσμα της έρευνας σε πραγματικές αλλαγές, ε, διότι η πραγματική πρόκληση είναι η εφαρμογή των πολιτικών και θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, ποιοι είναι οι καλύτεροι δυνατοί δείκτες ε, για την ε, ορθή εφαρμογή των πολιτικών, επόμενη διαφάνεια, να και το Μονρεάλ, έτσι θα είναι και του χρόνο ελπίζω να έρθετε όλοι. Και αν θέλετε να μάθετε και περισσότερα για τη Σύνοδο 11, ο Δόκτωρ Πίντο αύριο θα σας μιλήσει για το Μόντρεαλ και για τη Νέα Σύνοδο στην Ολομέλεια στις 9. Και η τελευταία διαφάνεια. Αυτή είναι η εταίροι μας ε, αύριο, οι βασικοί διοργανωτές ε, και έχουμε πάρα πολλούς εταίρους. Ευχαριστούμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπρε. Έχει ζητήσει το λόγο. Στη θέση 198. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάντηση αυτή για την ευκαιρία που μου δώσατε εκπροσωπώ μια νέα πρωτοβουλία η οποία λέγεται Gender Insight, Gender in Science. Το όραμά μας είναι ότι η αηφορία δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί αν πραγματικά το φύλλο και η επιστήμη, η προβληματική του φύλλου και η προβληματική της επιστήμης δεν συνδυαστούν. Πρέπει να πείσουμε λοιπόν αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν υπόψη τις διαστάσεις αυτές στις αναπτυξιακές τους πολιτικές. Νομίζω ότι αυτή εδώ η συνάντηση έχει προσφέρει πολλές και σημαντικές ιδέες. Και άκουσα και πολλές ριζοσπαστικές προτάσεις και επίσης ιδέες ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στην απλή συνεργασία και να περάσουμε σε δράση. Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό σημείο για όλα, τα, για όλα τις συναντήσεις κορυφής. Πρέπει να δούμε πέρα από τις διαπιστώσεις λοιπόν τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικά. Η συνάντηση αυτή νομίζω ότι θα το πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πια χρόνο για συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην Ελίζαμπεθ για να κλείσει τις εργασίες μας. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά μου Ολοκληρώνω αυτήν την ε, διάσκεψη. Τονίσαμε λοιπόν ότι η διάσκεψή μας έχει να κάνει με το φίλο με τους άνδρες και τις γυναίκες και την πολυμορφία που τους ε, διακρίνει. Και επίσης ασχοληθήκαμε με την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας, επιστημονική έρευνα η οποία πρέπει να γίνεται προς όφελος όλων των μελών της ε, κοινωνίας, ανδρών και γυναικών και όλων των κοινωνικών στρωμάτων, έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουν εξίσου τα ίδια ωφέλη, ακόμα και οι γυναίκες και οι υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Αυτό λοιπόν ήταν και ο στόχος της διάσκεψής μας. Η διάσκεψη για το φύλλο δεν είναι μόνο ένα συνέδριο, αλλά μια πρωτοβουλία για αλλαγή. Εσείς είστε κομμάτι λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που μας δώσατε, να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του και να κλείσω λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε τα πράγματα είναι η συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ελίζαμπεθ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Νομίζω πως πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει να αρχίσει η εκπαίδευση από το σχολείο. Πρέπει από το σχολείο, από μικρή ηλικία ήδη τα παιδιά να μαθαίνουν ότι είναι ίσα σε όλους του τομείς της ζωής τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτή η εκπαίδευση αρχίζει από την οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.